Ja, liebe Kolleginnen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, θα ήθελα θερμά να σας καλωσορίσω στην απογευματινή μας αυτή συνεδρίαση απόψε. Συνεδριάσαμε λίγο παραπάνω με τους συντονιστές και κάπως μετατέθηκε το πρόγραμμα και εξάλλου η αντιπρόεδρος κ. Μουσκαρντίνη βρίσκεται καθοδόν από το αεροδρόμιο προς το Ευρωκοινοβούλιο. Και ανταυτίσα ξεκινώ τη συνεδρίαση λοιπόν τώρα εγώ. Θα ήθελα πραγματικά με όλη μου την καρδιά να σας καλωσορίσω θερμά κυρία Υπουργέ για δεύτερη φορά εδώ ενώπιον μας μπροστά μας στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Θα έλεγα οι σχέσεις εργασίας αποδείχθηκαν πολύ καλές οι σχέσεις μας με την Δανέζικη Προεδρία του Συμβουλίου έτσι αναπτύχθηκαν πολύ θετικά. Και στον τομέα αυτό για το εμπόριο έχουμε δύο πολύ νομο... σημαντικές νομοθετικές προτάσεις υπό την πρωτοκαθεδρία του Συμβουλίου που μπόρεσαν να προαχθούν. Αφενός το θέμα των διμερών επενδύσεων, συμφωνιών επενδύσεων, όπου μετά από έντονες και μακρές διαπραγματεύσεις εκπονήθηκε ένας λογικός καλός συμβιβασμός και φυσικά και το θέμα του Γενικού Συστήματος Προτιμήσεων, δασμολογικών προτιμήσεων, όπου καταφέραμε και εκεί να ολοκληρώσουμε με θετικό τρόπο. Και θα έλεγα το ένα ή το άλλο θα ανταλλάξουμε ως απόψεις ε, επ' αυτών των θεμάτων. Για παράδειγμα για την εντολή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία διότι γνωρίζετε κυρία Υπουργέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την επιθυμία σε σχέση με την Ιαπωνία για την διαμόρφωση της εντολής να αναβληθεί αυτό το θέμα μέχρι ότου θα υπάρξει τοποθέτηση πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της Ιαπωνίας ώστε να ενταχθεί και αυτό στην εντολή όπως πρέπει με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό συνολικά παρακαλώ στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις να λαμβάνετε υπόψη και μόνο όταν το Κοινοβούλιο αντίστοιχα θα έχει ενημερωθεί και τοποθετηθεί να μπορεί να προχωρήσει κάτι. Διότι είναι φυσικό ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή στο τέλος της διαδικασίας να μπορούμε να εκφράζουμε την άποψή μας ως Ευρωβουλή. Και αν δεν λαμβάνεται πιο πριν υπόψη και απορρίπτουμε στο τέλος ως Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό θέλουμε όλοι να το αποφύγουμε φυσικά. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε, καλώς ήρθατε θερμά και θα ήθελα και τους συνεργάτες σας, γυναίκες και άνδρες, κυρίες και κυρίους, να ευχαριστήσω για τη συνεργασία, τη θετική συνεργασία των σχέσεων μεταξύ μας διότι μπορώ να φανταστώ δεν είναι καθόλου εύκολο για αυτές και για αυτούς να συνεργάζονται με το Κοινοβούλιο. Πολλές φορές δημιουργούνται τριβές. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και το επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας. Έχετε τον λόγο κυρία Υπουργέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω, νομίζω ότι είναι λυπηρό που δεν είναι εδώ ο κύριος ε, ε, Μορέιρα. Λυπούμε που δεν τον βλέπω εδώ και του εύχομαι καλή ανάρρωση. Καλωσορίζω λοιπόν την ε, συζήτηση αυτή ε, γιατί ε, είναι και απόρρια του εκδημοκρατισμού των θεσμικών οργάνων μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας. Η συνεργασία μας και θα συμφωνήσω με τον Πρόεδρο ήταν πραγματικά πολύ καλή και έδωσε κάποια δημοκρατικά αλλά και ορθά αποτελέσματα και προσωπικά να σας πω, σε προσωπικό τόνο, να σας πω ότι με μεγάλη ευχαρίστηση συνεργάστηκα μαζί σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την καλή συνεργασία. Κυρίως θα ήθελα να υπογραμμίσω την ε, σημασία των ε, αποφάσεων που πήραμε και των συμφωνιών που επιτύχαμε σε δύο ε, θέματα πολύ σημαντικά η πολιτική συμφωνία που επετέφθη πριν μερικές συμφωνίες ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων ε, αφορά και δύο κανονισμούς και είναι πρακτική απόδειξη της ε, καλής διοργανικής νομοθετικής συμφωνίας μέσα από συμφωνία, από διάλογο, από αμοιβαίες υποχωρήσεις καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ ικανοποιημένη ε, σχετικά με τους ε, δύο αυτούς κανονισμούς, λοιπόν, χαίρομαι που φτάσαμε σε αυτό το ε, θέμα. είναι τους δύο κανονισμούς και επομένως μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση για την περαιτέρω αύξηση του ε, εμπορίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας στο σύνολό του, αλλά βεβαίως τον κύριο Μορέιρα ακόμα ειδικότερα για τη συνεργασία. Και σας ε, υπόσχομαι ότι θα περάσω αυτή την καλή ε, εμπειρία της συνεργασίας με την Επιτροπή σας και στους Κυπρίους συναδέλφους, τους οποίους θα δώσουμε την σκητάλη. Οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να βοηθηθούν ε, από αυτά τα ε, μορομερή εμπορικά εργαλεία και ε, χαίρομαι και γιατί και στην, την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, Ολομέλεια υπήρξε ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά το ψήφισμα του εισηγητή όσον αφορά τώρα το σύστημα γενικευμένων προ, προτιμήσεων και εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εμπλεκόμενους για την πολύ καλή συνεργασία. Η συνεργασία μας είναι ζωτικής σημασίας, όχι μονάχα ε, στον καθορισμό ε, των ε, επιθετικών στάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις ε, ε, παρούσες ε, συνθήκες. Το προηγούμενο χρόνο, αλλά και από ό,τι φαίνεται το 2012, δεν θα έχουμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του εξωτερικού εμπορίου μπορούμε να έχουμε μια αύξηση 0,7% στο ΑΕΠ, άρα είναι σημαντικό το εξωτερικό εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν ε, δεν, είχαμε, αν δεν είχε ε, και την ε, ζήτηση του εξωτερικού εμπορίου θα βρίσκεται σε ύφεση Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο ε, σημαντικό είναι το θέμα αυτό και μην ξεχνούμε ότι εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Επικράτειας θα λάβουν χώρα τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης και για το 2012. 2% ε, του ΑΕΠ και 2 εκατομμύρια ε, θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έχουν σχέση με το εμπόριο. Οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης ε, βεβαίως ε, θα πρέπει στη διάσκεψη κορυφής ε, την 29η Ιουνίου να συζητήσουν τα θέματα αυτά. Και αυτό θα είναι πολύ θετικό, διότι υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι, εμπορικοί, οι εμπορικές οι εμπορικές συμφωνίες και το εμπόριο μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, και ε, υπό τις οδηγίες των Υπουργών Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν ε, την 31η Μαΐου. Μην ξεχνούμε επίσης ότι και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου μία ε, μακροτενής παράγραφος ασχολείται με το εμπόριο. Οι διαπραγματεύσεις, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ε, η διαπραγμάτευση μάλλον ε, για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνία ήταν κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Ολοκληρώθηκε η λεγόμενη scoping exercise και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την πραγματική συνεργασία. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά θετικά. Γνωρίζω βεβαίως τις ευαισθησίες που σχετίζονται με τις ε, Διαπραγματεύσει αυτές, αλλά να πω ότι και η προπαρασκευαστική εργασία που έγινε με την Ιαπωνία είναι η καλύτερη που έχει γίνει όσον αφορά την προετοιμασία οποιασδήποτε άλλη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Έχει δεσμευτεί πλήρως ε, η Ιαπωνία και εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσουμε τελικά να πούμε ένα ναι ή ένα όχι, αν ε, θα θέλουμε ή όχι να ξεκινήσουμε το δρόμο αυτό με την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι πολύ σκληρές. Ε, ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται τα μάλα για το ε, θέμα αυτό. Ε, ξέρει ποιες είναι οι πρόνοιες που προβλέπει το Συμβούλιο για τις διαπραγματεύσεις, ε, ξέρει τη θέση της Κομισιόν και πρέπει να σας πω ότι το Συμβούλιο με μεγάλη προσοχή περιμένει να ακούσει τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Είμαστε είμαστε δεσμευμένοι, στρατευμένοι στο θέμα της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ε, στις αγορές και επομένως θέλουμε και στις μεγάλες και στις μικρότερες ε, ε, χώρες να βελτιώσουμε την πρόσβαση που μπορούν να έχουν οι εταιρείες στην αγορά. Είδαμε ε, τις ε, προόδους ε, στις διαπραγματεύσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί για το FTA. Υπάρχουν πολλά ζητήματα προς επίλυση και ευελπιστούμε ότι τον, Ιούλ, τον Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Ε, το, οι συμφωνίες ε, στα πλαίσια και του ΠΟΕ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η, πρόσβαση, η, η ένταξη στην Ρωσία οπωσδήποτε θα είναι ένα καινούριο στοιχείο και θα μπορέσει να δώσει όθηση και στους δικούς μας εξαγωγείς αλλά και στους Ρώσους εξαγωγείς. Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία σύντομα θα είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμα ένα βήμα ε, ανοίγοντας εμπορικά κεφάλαια τα οποία θα ξεπερνούν τις δεσμεύσεις ε, του ΠΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη επίσης να ε, διευρύνει την οικονομική της συνεργασία με την Ρωσία. Δυστυχώς δεν είχαμε σημαντικές δεν είχαμε σημαντικά ανοίγματα όσον αφορά συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ξεπεράσουμε ε, όλες τις παλιές απόψεις όσον αφορά τον προστατευτισμό και να προχωρήσουμε σε ε, πραγματικό ελεύθερο εμπόριο. Είναι προφανές ότι και στο μέλλον θα προστατέψουμε ε, τα συμφέροντα των ε, εμπορευομένων μας ε, και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις για να το πετύχουμε αυτό οι διαπραγματεύσεις πιστεύουμε ότι μπορούν να ξεκινήσουν ε, και ανοίγοντας νέα κεφάλαια το δεύτερο ε, εξάμεινο του 2012. Και οι διατλαντικές συμφωνίες αποτέλεσαν προτεραιότητα για μας. Είχαμε καλή επαφή με τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα την ενδιάμεση επισκόπηση και μία πρώτη συνολική αξιολόγηση περί τα ε, τέλη του 2012. Υπάρχει δέσμευση και από τις δύο πλευρές για να δούμε πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ε, στη μεγαλύτερη από δημιουργία συστήματος FTA, στη μεγαλύτερη, λέω, εμπορική συμφωνία FTA. και θα θέλαμε να ε, ανοίξουν τα κεφάλαια αυτά ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως ε, στα πλαίσια αυτά θα ενδυναμωθεί και δεν θα αποδυναμωθεί ο ΠΟΕ και το σύστημα πολυμερών συμφωνιών. Ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τους ε, γείτονές μας ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με την Ουκρανία τώρα έχει γίνει η έκθεση αξιολόγησης και όσον αφορά τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις αρνητικές προς την, ε, όσον αφορά την Ουκρανία και δυσκολεύει η κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Ουκρανία να ξαναβρει το δρόμο των ευρωπαϊκών αξιών, αλλιώς θα είναι δύσκολη η κατάσταση με την Γεωργία, την Μολδαβία και την Αρμενία ε, προχωράμε με, τα, με τις συμφωνίες για FTAs και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις αυτές και έτσι ώστε οι τρεις αυτές χώρες να έχουν πλέον ε, ενσωμάτωση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είχαμε scoping exercises με την Ιορδανία, τον, το Μαρόκο και την Τινησία που θα ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτές ε, οι FTAs, αυτές οι συμφωνίες ελευθερών εμπορίου θα είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, για την περιοχή. Επίσης, ε, να σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη θα έχουν ολοκληρωθεί υπό δική μας Προεδρία και έχει αποφασιστεί να ξεκινήσουν τις ε, επόμενες, ε, ε, να ξεκινήσουν άμεσα και η απόφαση λήφθη τις προηγούμενες εβδομάδες, συνεργασία και διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ. Όσον αφορά τώρα την Κολομβία και το Περού, αργότερα αυτό το μήνα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Κολομβία και για το Περού γνωρίζουμε ότι και εσείς ε, προβληματίζετε όσον αφορά ε, την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελευθερού Εμπορίου με τις χώρες αυτές. θέλουμε κάποιες διασφαλίσεις και θέλουμε να γνωρίζουμε την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως ανησυχεί και εκφράζει την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν ε, οι διαπραγματεύσει αυτές και βεβαίω τα ζητήματα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αηφόρου ανάπτυξη είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, ε, Ε, υπάρχει ακόμα ένα προβληματικό πρωτόκολλο, είναι το ε, ε, πρωτόκολλο το οποίο ακόμα εκρεμεί τη συμφωνία για τα κλωστοφιδουργικά με το Ουσμπεκιστάν. Και εκεί ε, ε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο είναι ε, η υποχρεωτική εργασία των ανηλίκων στο Ουσμπεκιστάν και επομένως θα πρέπει με εποπτεία επιτόπου να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Όσον αφορά το Πακιστάν, ξέρουμε, το ξέρετε πώς είναι η κατάσταση, είναι πολλοί οι Πακιστανοί οι οποίοι υποφέρουν ως αποτέλεσμα των τρομερών πλημμυρών και γενικώ των φυσικών καταστροφών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσεις απέναντι στο Πακιστάν. Ε, έχει κάνει προτάσεις ε, το Συμβούλιο ε, και στο πρώτο τριμερή διάλογο το Συμβούλιο υπέβαλε κάποιες συμβαστικές προτάσεις και ευελπιστούμε ότι σύντομα ε, θα έρθουμε σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Θέλει το Συμβούλιο να κλείσει το φάκελο αυτό. Επανερχόμενοι στην προσπάθειά μας ε, για να ανοίξουμε τις αγορές, ε, να κάνουμε σωστό ανταγωνισμό, πρέπει να πω ότι αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία ανάπτυξης. Ελεύθερη πρόσβαση ε, στην αγορά δημοσίων προμηθειών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων χωρών. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία ε, κάνοντας κάποιες πρώτες προτάσεις υπό δική μας προεδρία. να σας πω και δύο λόγια όσον αφορά το Regional Marketing, το οποίο συζητιέται εδώ και αρκετό καιρό. Ε, σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο μετά την πρόταση της Επιτροπής του 2005. Όμως, η μεγάλη στήριξη του Κοινοβουλίου για, προς τον κανονισμό διευκόλυνε τη συζήτηση στο Συμβούλιο όπου η πλειοψηφία των μελών εξέφρασαν την βούληση για νέα επικοδομητική προσέγγιση ε, μιας νέας ε, πρότασης της ε, Κομισιόν. Όμως ε, η Κομισιόν δεν έχει ακόμα υποβάλει ε, τέτοια πρόταση όσον αφορά την άκτα. Ε, λαμβάνουμε υπόψη, είναι τις τελευταίες εξελίξεις. Το Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο, μάλλον η Κομισιόν, ζήτησε νομική γνωμοδότηση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, σύμφωνα με το θεμελιώδη, τις θεμελιώδεις αρχές Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΟΕ ε, και η αποφάση του είναι πάρα πολύ ε, σημαντικός για τις εξελίξεις στο εμπόριο. Στη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας είχαμε νέες προσεγγίσεις ε, στην Γενέβη όσον αφορά ζητήματα τα οποία είχαν φτάσει ε, σε ε, νεκρό σημείο και σε αδιέξοδα. Αυτά δεν είναι καθόλου εύκολα πράγματα γιατί υπάρχουν πολλά μέλη του ΠΟΕ που δεν θέλουν να μετακινηθούν από τις ε, θέσεις τους. Εμείς ε, προσπαθούμε να ε, ξεπεράσουμε προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη ειδικά ζητήματα όπως είναι ας πούμε οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες κτλ. να σας πω, ο, ο, να σας πω ότι ε, η trade facilitation μπορεί να αποτελέσει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ΠΟΕ. Επίσης, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ανοίξει συζήτηση και για άλλα κεφάλαια, όπως ας πούμε είναι η πολυμερής πρόσβαση στις υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως, μην ξεχνούμε ότι είναι, αν όχι ο σπουδαιότερος, ένας από τους σπουδαιότερους εμπορικούς εταίρους των περισσότερων αναπτυσσομένων ε, χωρών. Επομένως γίνεται μια προσπάθεια να εξευρεθούν συμφωνίες ε, ε, όσον αφορά την νέα, τα νέα, τις νέες συμφωνίες για το καθεστώς γενικευμένων προτιμήσεων. μετά την ε, θέση ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, έγινε μια, μια διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου έτσι ώστε να ξεκινήσουν καλύτερα οι διαδικασίες αυτές και ασχοληθήκαμε κυρίως με τις πιο τροτές, πιο ευάλωτες χώρες. Επίσης, απελευθέρωση πράσινου εμπορίου και αυτό ε, ξανά ήρθε ε, στο τραπέζι μετά από το 2009. Μετά από έτοιμα της ε, διάσκεψης των Υπουργών, του Συμβουλίου συγγνώμη, των Υπουργών Εξωτερικών την 6η Μαΐου ε, έλαβε χώρα και Συμβούλιο των Υπουργών ε, Εμπορίου την 31η Μαΐου. Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι δυνατές ε, κατευθύνσεις. Όμως μπορώ να σας πω ότι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που ακούστηκαν ήταν οι πολυμερείς συμφωνίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ε, που οδήγησαν σε πρωτοβουλίες όπως η ΣΥΤΑ ας πούμε. Νομίζω ότι πρόκειται για ε, θέματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν ε, περαιτέρω. Επίσης και μέσω της ΕΠΙΚ μπορούν να γίνουν περαιτέρω διεργασίες. Βεβαίως ξέρουμε ότι η ε, πρόκληση είναι ε, μεγάλη έτσι ώστε να έχουμε την απαραίτητη στήριξη μιας κρίσιμης μάζας εμπορευμένων έτσι, και χωρών. Ε, αυτό άλλωστε αποτελεί και αντικείμενο του διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Τέλος, να σας πω ότι ήταν μεγάλη χαρά να ασχοληθώ με αυτή την πολύ σκληρή δουλειά και με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Συνεργασία και με την Κομισιόν και με εσά ήταν εξαιρετικά ε, ενδιαφέρουσα. Θα ολοκληρωθεί σύντομα βεβαίω η εμπειρία αυτή, αλλά είμαι σίγουρη ότι και ε, οι ε, συνάδελφοι που θα πάρουν τη σκητάλη από εμά με τη δικιά σας καλή επαφή και συνεργασία θα ολοκληρώσουν και, και άλλους Ευχαριστώ. Ja, ganz herzlichen Dank. Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την σφαιρική επισκόπηση που μας δώσατε συνολικά για τα θέματα που συνδιαμορφώσατε και έχετε προαγάγει. Τώρα θα έχουν οι συνάδελφοι την δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και περωτήσεις. Ο πρώτος γύρος νομίζω έχει ήδη ολοκληρωθεί στον κατάλογο. Αντία Μάρτιν, οι τρεις δεν έχουν ζητήσει άλλοι τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τα λόγια σας, για τις πληροφορίες που μας δώσατε, για την καλή σας διάθεση σε όλη τη διάρκεια της Προεδρίας για να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο. Και να σας συγχαρώ και για μερικές πρόοδους που, μπορέσαμε να έχουμε σε αυτήν την Επιτροπή. Δύο ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες. Η μία που αφορά στην ε, υπερδραντική συνεργασία. Εσείς είπατε ότι προχώρησε και θέλω να παρακαλέσω, θα μπορούσατε να μας ε, πείτε προκαταβολικά αν τίνουμε προς μία συνολική συμφωνία ή απλώς έχουμε θέματα στα οποία συμφωνούμε παραπάνω, οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε μερικές συμφωνίες. Δεύτερη ερώτηση σχετικά με το ΑΚΤΑ. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο είχε ένα σωρό ακριάσεις, ακροάσεις, συνεδριάσεις όλους τους, με, με όλους τους κλάδους. Ένα από τα θέματα που διαφάνηκε σε αυτές τις συνεδριάσεις ήταν η ερώτηση. Μα σας πέρασε ποτέ από το νου να προτείνετε ένα ευρωπαϊκό άκτα και για να μην πάω και πιο μακριά, δηλαδή σήμερα είχα επισκέπτες και μου κάνανε αυτή την ερώτηση. Τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Άκτα, μία πρόταση της Κομισιόν που να φύγει αυτά τα θέματα. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε ο Πρόεδρος και η Επιτροπή σας. Υπήρξε πνεύμα συνεργασίας και συμβιβασμών με την Προεδρία και το χαιρετίζουμε αυτό. Επίσης και για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα θέματα ανάπτυξης πολύ σημαντικά για μένα και την ομάδα μου. Επίσης θέλω να καλωσορίσω, όχι να καλωσορίσω, να σας συγχαρώ. Να σας συγχαρώ επίσης για το πνεύμα που καταδείξατε σε σχέση με το ζήτημα του Πακιστάν. Λοιπόν, έχω κάποιες μικρές ερωτήσεις να διατυπώσω. Είπατε ότι για το θέμα της Ιαπωνίας θα μπορούσατε να φανταστείτε ή θα θέλατε να δείτε να εμπλέκετε περισσότερο το κοινοβούλιο από ό,τι στο παρελθόν. Ωραία είναι να το ακούει κανείς αυτό. Έχουμε προβλήματα και στο τέλος μπορούμε να εγκρίνουμε ή να καταψηφίσουμε και δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό αυτό. Γίνονται ήδη κάποιες σκέψεις για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η εμπλοκή του Κοινοβουλίου και σε σχέση με την εντολή και το πλαίσιο της εντολής. Ή δεν, έχει, δεν μπορεί να γίνει ακόμα αυτό δεκτό από το Συμβούλιο. Και για το Ουσμπεκιστάν που αναφέρατε επίσης όπου το Κοινοβούλιο έθεσε όρους και προϋποθέσεις δεν ξέρω, ίσως και αυτό θα μπορούσε να ήταν μια δυνατότητα και για άλλες περιπτώσεις άλλων χωρών. Συζητήσεις γίνονται στο Συμβούλιο για κάτι τέτοιο. Πώς αυτό θα μπορούσε να είναι μια βάση θεμέλιο εργασίας. Μετά αναφερθήκατε στο θέμα των ε, ΣΕΤΑ, διαπραγματεύσεων ΣΕΤΑ. Ασκήθηκαν επικρίσεις από τα κράτη-μέλη ότι δεν είχαν ενημερωθεί καλά και διαρωτώ με, με ποιο τρόπο το Συμβούλιο στοχεύει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει το θέμα των διαπραγματεύσεων ΣΕΤΑ και πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές τις διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κύριος Μάρτιν τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Καλύψατε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και θα ήθελα τρία από αυτά να επιλέξω. Πρώτον, οι νομικές μας υπηρεσίες εξέτασαν κάποιες από τις διαδικασίες συναπόφασης που μας έχουν υποβληθεί από το Συμβούλιο Προτάσεις για την Κολομβία, Νότια Αμερικής και για τη Συμφωνία ΕΕ Ρωσίας. Σύμφωνα με τη νομική αυτή τους νομομαθείς και σύμφωνα με τις απόψεις μας εμπεριέχουν κάποια ναι, διαδικασίες συνενετικές ε, και από πλευρά της ε, αξιολόγησης ε, είπαν ότι υπάρχουν πτυχές που πρέπει να εξετάσουμε όσον αφορά τη συναπόφαση και αυτό σε σχέση με τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο μέλλον να μας αποστέλετε μόνο τότε συμφωνίες προς έγκριση όταν θα εντάσσονται πλήρως στην συναπόφαση και στις διαδικασίες συναπόφασης και να εξευρεθούν λύσεις ε, για τα προβλήματα. Δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση το κοινοβούλιο να παρακάμπτεται και να λέμε μόνο ναι όχι να δεχόμαστε να απορρίπτουμε κάτι ενώ έχουμε δικαιώματα συναπόφασης και τροποποίησης. Δεύτερη ερώτηση. Δεν στοχεύει τόσο πολύ στην Δανία, στην ίδια την Δανέζικη Προεδρία, αλλά περισσότερο γενικότερα στο Συμβούλιο. Γίνονται συζητήσεις σοβαρές και σε βάθος για την αντιστοιχία σε σχέση με την αντιμετώπιση χωρών, όπως αναφέρατε, παράδειγμα την Ουκρανία. Ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά, από το Συμβούλιο είχαμε την αναβάθμιση σε σχέση με τη Συμφωνία για το Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν μια χώρα που εκμεταλλεύεται τα παιδιά, που ε, ε, έχει την υποκατοχή τη λωρίδα της Γάζας ε, και την δυτική Όφθη και έχουμε εμπορικές σχέσεις με μια τέτοια χώρα. Ταυτόχρονα όμως για την Ουκρανία που συμφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα, παγώνουμε τη συνεργασία μας. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ε, συνέπεια και συνεκτικότητα και μετά τα όσα είπατε για την πολιτική, για την ανάπτυξη θετικά τα αντιμετωπίζω. Όμως είχαμε και τον, ε, την τροποποίηση του κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά που θα αποκλείσει την δυνατότητα πρόσβασης προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες, χώρες στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν όλα αυτά συνάδουν μεταξύ τους. Εσείς παρακαλώ συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ Θέλω πρώτα να ξεκινήσω, λέει ο κύριος Σόλτς, Υπουργέ, για το ότι μας αναφερθήκατε σε ένα ευρύ φάσμα όσον αφορά τις προσπάθειες που γίνονται να προαχθούν αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας της Δανίας στο Συμβούλιο για τα θέματα τα εμπορικά του εμπορίου. Άκουσα προσεκτικά τον μεγάλο κατάλογο των μερικών επιτευγμάτων, εν μέρη επιτευγμάτων, το, του συνεχιζόμενου έργου και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Φυσικά θα δοθεί σκητάλη από την Δανέζικη Προεδρία, φυσικά στην επόμενη Προεδρία. Και η Κοινοβουλευτική μας ε, Επιτροπή θα υποστηρίξει αυτή την ε, αλληλουχία πραγμάτων σε σχέση με την επόμενη Προεδρία. Άκουσα επίσης αυτό το οποίο είπατε για τη στενή διασύνδεση μεταξύ δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης και του ρόλου του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών θεμάτων. Ερώτηση, ποιες συγκεκριμένες προτάσεις μπορείτε εσείς να μας αναφέρετε ότι θα εξετάσει η Προεδρία και θα υποβάλει, θα, θα καταθέσει η Προεδρία ως συνεισφορά κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας για αυτά τα θέματα, επανερχόμενος φυσικά στη δήλωσή σας ε, ως κύρια πρόκληση για την εμπορική συνεργασία για την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση και των κλιματικών αλλαγών και προκλήσεων. Αναφέρατε την προσπάθεια, τη Διεθνή Συμφωνία για το πράσινο εμπόριο, Green Trade. Έχω κάποιες ιδέες και απόψεις, αλλά επανερχόμενος σε αυτό που είπατε πιο πριν, για τις ε, σχέσεις μας με τις ε, ΗΠΑ, δηλαδή ΕΕ Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, διατλαντική συνεργασία, με οδηγεί στη συνάφεια, στη διασύνδεση τη ερώτηση πώ θα αντιμετωπίζατε τι προσπάθειε ε, των ΗΠΑ το 2020 να είναι η υπερδύναμη στην παραγωγή ενέργειας, αυξάνοντας την παραγωγή ενέργειας και πηγών κατά 20% περισσότερο σε σχέση με το σημερινό επίπεδο και ταυτόχρονα μειώνοντας τις τιμές για τις ε, θερμικές μονάδες ε, του αερίου, των ε, εκπομπών για, το αέ, για τα αέρια του θερμοκηπίου σε σημαντικό βαθμό. Τι γίνεται σε σχέση με την Ευρώπη όταν έχουμε 2,35 δολάρια και θα έχουμε διαφορετικές τιμές και για την Ασία και άλλους. Αυτό θα οδηγούσε στον κίνδυνο αυτός ο ανταγωνισμός με βάση αυτό το συγκεκριμένο πεδίο να στοχεύει ή να είναι επικίνδυνο να στοχεύει αυτή την πράσινη, αυτό το πράσινο εμπόριο που θέλουμε να ευδοκιμήσει και να πετύχουμε. Πώς θα το αντιμετωπίζατε αυτό. Και σε σχέση με το ε, εγχείρημα ε, ITT για την ε, διάσκεψη κορυφής Ρίο 20 χρόνια μετά από την πρώτη συμφωνία. Τι μπορεί να γίνει σε σχέση με διεθνείς συμφωνίες για να αποφύγουμε την αποψήλωση του τροπικού δάσους, να μην συνεχιστεί δηλαδή η υλοτομία και καταστροφή των τροπικών δασών ε, της Αμαζονίας. Πώς θα υποστηρίζατε αυτούς τους στόχους ε, στην διάσκεψη κορυφής Ρίο μετά από 20 χρόνια, Ρίο συν 20. Μετά, αναφερθήκατε στις προκλήσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου υπό το δικό σας πρίσμα νομικά και όλων των θεμάτων που εμπλέκονται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις και όλους τους εμπλεκόμενους στο διεθνές εμπόριο οι δικές σας προτάσεις ποιες είναι και πώς διαμορφώνονται για να ξεφύγουμε, να διαφύγουμε από το αδιέξοδο του γύρου διαπραγματεύσεων της Ντόχα. Ίσως θα μπορούσε πολυμερός να γίνει κάτι για να βρεθεί μια λύση. Βλέπετε μια λύση να διαμορφώνεται συγκεκριμένα με κάποια προοπτική για να μπορέσει να ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Ολοκληρώνω εδώ να μην μακρηγορήσω. Ευχαριστώ. Καλύτερα ναι που ολοκληρώνεται εδώ. Δύο παρεμβάσεις τώρα. Οι δύο που ακολουθούν και μετά θα λάβει τον λόγο Υπουργό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά δεν θα μακρηγορήσω. Έχω συγκεκριμένες εξειδικευμένες ερωτήσεις. Θέλω να εκτιμήσω θετικά το θετικό πνεύμα και την θετική διάθεση της ε, Δανέζικης Προεδρίας για την ανάπτυξη προαγωγή των θεμάτων του διεθνούς εμπορίου που εμπειρικά κιόλα όσον αφορά μια παραδοσιακά εξαγωγό χώρα που αντιμετωπίζει τα θέματα του διεθνούς εμπορίου με ιδιαίτερη ευαισθησία και ως ιδιαίτερη σημασίας και σπουδαιότητας για την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε θετικά. Επίσης έπρεπε να αντιμετωπίσετε πολλά περίπλοκα θέματα και θέματα τα οποία πρέπει πραγματικά να υπογραμμιστούν μεταξύ αυτών πέρα από κάποιες διεργασίες scoping διαπραγματεύσεις ε, με κάποιες ε, τρίτες χώρες ε, και συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά. Θέλω να τονίσω ένα εξειδικευμένο θέμα για τις συμφωνίες διμερούς, διμερών επενδύσεων, διμερείς συμφωνίες επενδύσεων. Μπορώ να σας ευχηθώ λοιπόν κάθε επιτυχία στην τελευταία φάση, τις τελευταίες ημέρες της Προεδρίας σας και θέλω να ευχαριστήσω για όσα κάνατε κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της Προεδρίας σας πιο πριν. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, αυτά είχα να δεν ασκήθηκαν επικρίσεις, ωραίο αυτό καμιά φορά να το βλέπει κανείς και να το ακούει. Ο κύριος Στάσνη παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νόμιζα ότι το όνομά μου είναι Άραντιλ, αλλά Έστω Στάσνη. Και εγώ θα είμαι σύντομος και ευχαριστώ την Δανέζικη Προεδρία και την Υπουργό ιδιαίτερα για το θετικό έργο το οποίο επιτελέσατε και την θετική προσέγγιση σας και την επιτυχή ε, έκβαση. Είχα κάποιες ε, ερωτήσεις για το ΙΤΑ και ανέμενα τώρα υπομονετικά για τις απόψεις και την τελική σας αξιολόγηση για αυτό το θέμα το ΙΠΑΣ είχε υπογραφεί μια συμφωνία πρόσφατα και για την ε, προσπάθεια που έγινε με τις χώρες της Αφρικής ε, σε Χέλες, Μαδαγασκάρι και κάποιες άλλες χώρες και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο ρυθμός των εξελίξεων θα επιταχυνθεί, θα επιβραδυνθεί τι πιστεύετε, τώρα που θα σταματήσετε να είσαστε προεδρεύουσα, μπορείτε να είσαστε ειλικρινείς μαζί μας και να μας τα πείτε ξεκάθαρα και στα ίσια. Τι πιστεύετε λοιπόν σε σχέση με αυτά. Αναμένω να ακούσω την άποψή σας. Και αυτό είναι προτέρημα υπό το πρίσμα αυτό να ξεφύγει κανείς από το αξίωμα της προεδρεύουσας και να μπορεί να μιλήσει πιο ελεύθερα και πιο ανοιχτά. Έχετε τον λόγο κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και πρώτα απ' όλα Κουτσέτ το όνομά σας Μπαντία ή Κουτσέτ μάλιστα πολύ σωστά λοιπόν για την διατλαντική εμπορική σχέση, εταιρική σχέση. Πιστεύω ότι είδαμε ότι υπάρχει μια προθυμία και από τις δύο πλευρές να υπάρξει κίνηση προς τα εμπρός, μια πρόοδος. Τώρα για το ότι θα πρέπει να είναι μια βαθύτερη, ευρύτερη συμφωνία από πλευρά του Συμβουλίου, λένε οι Ηνωμένε Πολιτείε ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοπλαίσιο γιατί διαφορετικά θα υπάρξει ένας νέος γύρος τύπου Ντόχα του ΠΟΕ, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και δεν νομίζω να ε, θέλει να γίνει κάτι τέτοιο κάποιο εμπλεκόμενο μέρος. Τώρα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις είναι σημαντικό θα έλεγα να βρεθούμε σε υψηλές προδιαγραφές για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και αυτές οι, υψηλού επίπεδου αναβαθμισμένες προδιαγραφές και ρήτρε να ισχύουν. Και τώρα, σε σχέση με τις συζητήσεις που συνεχίζονται, υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές να ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια. Για την άκτα, θα ήθελα να πω, δεν ήταν το πιο εύκολο θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας αυτό. Και αυτό είναι μάλλον εφημισμός κιόλα. Θα ήθελα να δω τι θα κάνει το Κοινοβούλιο αύριο και πώς θα διαμορφωθεί η απόφαση από πλευράς του Συμβουλίου. Αυτό που θέλαμε να δούμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και φυσικά νωρίς είχε πει το Ευρωκοινοβούλιο ότι θα ενδιαφερόταν να δει αν το Ευρωδικαστήριο θα ε, κατέβαζε τον πύχη όσον αφορά τα δικαιώματα σε σχέση με την χάρτα των δικαιωμάτων. Τώρα θα πρέπει να δούμε Πώς θα μπορέσει, πώς θα τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σημειώνουμε όμως τις απόψεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το αιρετό όργανο των πολιτών που ε, εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά αυτά που θα πείτε αύριο και σημειώνουμε καλώς ε, τις απόψεις σας. Στην κυρία Κέλλερ τώρα, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους σας για τα καλά σας λόγια, για την Ιαπωνία που αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι να δώσει μια εντολή. Είναι σαφές ότι συνταγματικά είναι ρόλος ε, του Συμβουλίου να θρώσει, να διατυπώσει μια τέτοια εντολή που θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την εντολή προχωρά. Όμως είναι σημαντικό να έχουμε χρόνο να ακούσουμε ο ένας τον άλλον και να, να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και είναι επίσης χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διεξαγάγει αυτές τις συζητήσεις σχετικά το Σεπτέμβριο, διότι μια γόνιμη συζήτηση και συνεισφορά του Κοινοβουλίου θα έχει επιπτώσεις για την αναβαθμισμένη ποιότητα της εντολής. Έχοντας αυτές τις άτυπες συζητήσεις και έχοντας το Κοινοβούλιο που υποβάλλει και αποστέλει προτάσεις και ιδέες ποιες είναι οι απόψεις του, Γνωρίζω ότι το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη αυτές τις απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου λαμβάνοντας την απόφαση υστερότερα. Δεν θέλω με κανένα τρόπο να υπάρξει αλλαγή τροποποίηση της συνταγματικής βάσης. Το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο θα δράσει, όμως με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα εισακούγεται και το Κοινοβούλιο. Τώρα για την ΣΕΤΑ, ΣΥΤΑ, Είχαμε μία συζήτηση στο, στην πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου στις 16 Μαρτίου και άτυπε συζητήσεις στο Συμβούλιο ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει ένα έγγραφο εναλλακτικών λύσεων και δυνατοτήτων για τη συνάντηση του Μαΐου. Συνέταξε λοιπόν ένα τέτοιο έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαμε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης πώς να, θα μπορούσαν να προαχθούν αυτά τα θέματα και σημειώσαμε και είπαν κράτη-μέλη ότι ενδιαφέρονται να υπάρξει απελευθέρωση, φιλελευθεροποίηση του πλαισίου για το πράσινο εμπόριο, green trade. Υπάρχουν πολλές προτάσεις ε, και νομίζω μπορούν να συνεισφέρουν με το να υπάρξει ένα νέο πνεύμα, νέες προτάσεις, νοπές ε, ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε σχέση με την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών από τον ΠΟΕ. Σε σχέση με το 2001 πολλές αναπτυσσόμενες χώρες πίστευαν ότι οι πλούσιες χώρες θα επέβαλαν στις αναπτυσσόμενες χώρες τι θα έπρεπε να κάνουν στη διάθεση και εμπορία των προϊόντων τους. Τώρα όμως είναι τα αναπτυσσόμενα, οι αναπτυσσόμενες χώρες, εκείνες οι οποίες αναγνωρίζουν την φιλοπεριβαλλοντική πτυχή Κένια, Κίνα, Ινδία, την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όταν βλέπουμε ότι ε, σε σχέση με ε, διάφορα προϊόντα θα υπήρχε ενδιαφέρον για το ελεύθερο ε, και πράσινο εμπόριο. Προτού δημιουργηθεί ένα πλαίσιο λοιπόν, έχουμε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και το βρίσκουμε πραγματικά γόνιμο, καρποφόρο αυτό το εγχείρημα και μπορεί και το Κοινοβούλιο να υποβάλει προτάσεις και είναι μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο έτσι. Τώρα για τα όσα είπε ο κύριος Μάρτιν. Μάλιστα, διάβασα αυτή την επιστολή του καθηγητή ε, και είδα την επιστολή αυτή εχθές το βράδυ. Και εχθές το βράδυ συνέταξα και μία απάντηση σε αυτή την ε, τοποθέτηση. Πολύ προσεκτικά μελετούμε και εξετάζουμε τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή. Τα παίρνουμε όλα πολύ σοβαρά, με σοβαρότητα τα αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνοντας λόγο για καλές προθέσεις, το Συμβούλιο αποφάσισε να επανεξετάσει την απόφαση για να ολοκληρωθεί να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σε σχέση με τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής. Θα τα κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καθυστερήσει η υπογραφή της συμφωνίας κατά τα τέλη αυτού του μήνα. Αλλά θα επανεξετάσουμε αυτά τα θέματα. Σε σχέση με τη συνεκτικότητα και συνοχή της πολιτικής μας, συμφωνώ μαζί σας να διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και συνέχεια της πολιτικής και συνοχή της πολιτικής πρέπει να γίνεται αυτό σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Έγιναν συζητήσει στο Συμβούλιο και με την περίπτωση συζήτηση τη Ουκρανία, αλλά και σε άλλα θέματα, όταν τα κράτη-μέλη αναφέρουν, για παράδειγμα, ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αν όλα αυτά λοιπόν θέτουν, είναι, ας το πω έτσι, κάποια κάποιο κίνητρο ή ε, μια δυνατότητα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν έτσι αυτό πρέπει να διασφαλίζεται για τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες. Πολύ προσέξαμε και επικεντρωθήκαμε στους κανονισμούς. Αυτές οι χώρες, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, που είναι οι πιο ευάλωτες να προσεχθούν ιδιαίτερα. Είναι δικό μας καθήκον και είναι στα χέρια μας να βοηθήσουμε για την ανάπτυξη αυτών των χωρών και πρέπει με τον κανονισμό και τις, ε, τους κανόνες που θα θεσπίσουμε να προαγάγουμε. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη υπουργό Περιβάλλοντος τώρα. Θα ήθελα όμως κάποια από τα θέματα για το Ρίο που αναφέρατε να, το, να τα καλύψω. Το Ρίο μετά από 20 χρόνια, Ρίο συν 20, διεξάγεται αυτή τη στιγμή ως διάσκεψη κορυφής στη Βραζιλία και για τις παραγράφους για το εμπόριο επικεντρωνόμενοι σε αυτά θέλουμε να δούμε πώς οι αναπτυσσόμενες χώρες μέσω του εμπορίου μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στη διάθεση των προϊόντων τους στις αγορές και να διασφαλίσουμε ότι το εμπόριο θα δρά υπέρ της αηφορίας στην ανάπτυξη, της βιώσιμης ανάπτυξης και με μεγαλύτερη ισότητα με πιο ισοδίκαιο τρόπο να αντιμετωπίζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες και τα προϊόντα τους. Τώρα, για το άλλο θέμα που είπατε δεν μπορώ να απαντήσω. Θα διαβιβάσω τις παρατηρήσεις σας στην Υπουργό Περιβάλλοντος που βρίσκεται στο Ρίο αυτή τη στιγμή και όταν επανέλθει τότε ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια τοποθέτηση. Ιδιαίτερα η διπλωματία και όσον αφορά και τις επαφές αυτές και την α, ε, ε, ανταλλαγή ερωτήσεων-απαντήσεων νομίζω μπορεί να λειτουργεί. Θα έλεγα ότι σε σχέση με τη Ουάσιγκτον, πρόσφατα επισκέφθηκα την Ουάσιγκτον και είχα συζητήσεις με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης Ομπάμα. Παρατήρησα και είδα ότι ενδιαφέρονται πολλοί αξιωματούχοι τον είπα, για το πράσινο εμπόριο. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση για την μείωση των ε, δασμών ε, στο επίπεδο του 5% με φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση. Οι ΙΠΑ έχουν συζήτηση για την εσωτερική, τον εσωτερικό ανεφοδιασμό τους και κάλυψη των ε, δικών τους ενεργειακών αναγκών εσωτερικά με τα μέτρα τα οποία ε, θα λάβουν. Ήταν ιδιαίτερα, είχε ιδιαίτερη προτεραιότητα στο θεματολόγιο στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα και στο Κογκρέσο και οι Δημοκράτες και οι Ρεπουμπλικανοί έχοντας εγγράψει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη είπαν και ότι πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία όσον αφορά την εισαγωγή εισαγόμενων προϊόντων, ενεργειακών προϊόντων ή πρώτων υλών για το γύρο της ΔΟΧΑ. Πώς μπορεί κανείς να προχωρήσει αν έχετε κάποιες ιδέες, οποιασδήποτε ιδέες ή προτάσεις. Κάτι που μπορεί να μην γνωρίζω, αδειμονώ να ακούσω τις απόψεις σας, διότι ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε ποιες είναι οι οποιασδήποτε προτάσεις σας για να προχωρήσουμε στο γύρο της Ντόχα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν αντιμετωπίζει αδιέξοδο. Ο γύρος διαπραγματεύσεων της Ντόχα έχει καταλήξει σε κάποια θέματα σε αδιέξοδο και προσπαθούν να δράσουν τα κράτη-μέλη ακόμα και σε μια χρονική στιγμή λόγω της κρίσης όταν υπάρχει πνεύμα προστατευτισμού, protectionism, υπάρχει η αντίστοιχη, το αντίστοιχο πλαίσιο από τον ΠΟΕ και μέσα από τον ΠΟΕ πρέπει να διασφαλιστούν περαιτέρω πρόοδοι για, το εμπόριο. Δεν ανησυχώ για ε, τα θέματα του ΠΟΕ, αλλά και για η λέσχη των 20, 20 αναγνώρισε τη σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων, αλλά δυστυχώς δεν, ανα, δεν ανέφερε τον γύρο της Ντόχα. Δημιουργούνται ανησυχίες πολλές φορές έτσι. Βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. λιμνάζουν τα πράγματα, έχουν αποτελματωθεί. Ας το πούμε και ας το ομολογήσουμε αυτό σε σχέση με τον γύρο της Ντόχα. Αλλά η πρόοδος ε, και το κλειδί για την πρόοδο είναι στα χέρια των ήπα και της Κίνας και πρέπει έτσι να εξεταστεί το θεματολόγιο των ζητημάτων του γύρου της Δόχα Είναι στα χέρια τους το κλειδί. Κύριε Στάσνη, σας ευχαριστώ πολύ για τα κολακευτικά σας σχόλια, τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ και για την ΣΥΤΑ. Ελπίζω ότι τα όσα είπα απαντούν και καλύπτουν την παρέμβασή σας. Τώρα, ακριβώς ε, λόγω των αφρικανικών αυτών ε, προσπαθειών υπάρχει μια όθηση να σημειωθεί πρόοδος. Θα σημειωθεί, θα γίνει ένας τριμερής ε, διάλογος, μια τριμερής διαπραγμάτευση για τα θέματα πρόσβασης στην αγορά. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει και κάποια ασφάλεια για τις χώρες EPA. Είναι δύσκολο όμως να προδικάσει κανείς αυτά που θα γίνουν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο να προδικάσει κανείς τι θα γίνει στο μέλλον και να τα προβλέψει όλα αυτά αλλά όλοι συμφωνούμε ότι αν το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι τόσο καλό και οι σχέσεις μας θα είναι τόσο θετικές όσο υπό τη δική σας Προεδρία θα έχουμε κερδίσει τη μάχη και τον αγώνα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι για τις επόμενες Προεδρίες θα είναι ένα θετικό παράδειγμα, ένα υπόδειγμα η δική σας Προεδρία πολλά θέματα προόδευσαν και προήχθησαν. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη Δανία. Ευχαριστώ. Ja, Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα ξεκινάμε με το επόμενο τμήμα της συνεδρίασής μας και πρόκειται τώρα σε σχέση με αυτό για μια ακρόαση για τις δυνατότητες που ανοίγονται, διανοίγονται να υπάρχει πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κεφάλαια για τα κεφάλαια όσον αφορά τη διεθνοποίηση. Δεν είναι κάποιο μυστικό βλέπετε ότι όλο και περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές εμπόριο αντιμετωπίζουν παγκόσμιο ανταγωνισμό και πρέπει να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό. Ιδιαίτερα σε, κρίσεις, σε περίοδους κρίσης η πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια είναι ουσιώδους σημασίας για την επιβίωσή τους. Και αυτό οδήγησε και στην ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που συντάχθηκε από πλευρά συναδέλφου μας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό οι δυνατότητες ε, να εξεταστούν πολύπλευρα, να δούμε πολύπλευρα ποιες δυνατότητες διανοίγονται. Και χαίρομαι ότι πραγματικά έχουμε μια ολόκληρη σειρά πραγματογνωμόνων, εμπαϊόντων, ώστε μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα και να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε η διαδικασία παγκοσμιοποίησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαμορφώνεται με επαρκή κεφάλαια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτα θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Κιούγι Ήτο που είναι από πλευράς ε, του ΟΑΣΑ, του ΟΣΑ για το Κέντρο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα υπεύθυνο για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην δική μας Επιτροπή. Έχετε αμέσω τον λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chair. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω όλους σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που έχω να κάνω την παρουσίαση αυτή. Είναι ε, σημαντικό να σας πω ότι εμείς σαν όσα έχουμε κάνει ε, μελέτες όσον αφορά το θέμα αυτό. Εγώ είμαι ε, υπεύθυνος για το ε, project. Μπορώ βεβαίως να σας δώσω να σας ε, δώσω τα αποτελέσματα αυτής ε, της ε, έρευνας. Αλλά αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω σήμερα είναι να κάνω μια επισκόπηση της έρευνας αυτής. Okay, so, uh, first, let me start... Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για το πρόγραμμα αυτό, το project αυτό. Το ξεκινήσαμε πέρσι. και βεβαίως ε, ε, βασίζεται στο ενδιαφέρον των ε, χωρών μελών. Όλες οι χώρες μέλη μας θέλουν να ενθαρρύνουν τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και βεβαίως προσπαθήσαμε να δούμε τα ενδιαφέροντα των χωρών μελών ε, να ταυτοποιήσουμε επίσης ποιε είναι οι αγορές στόχοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, να προωθήσουμε κάποιες ε, ιδέες οι οποίες είναι πιο σημαντικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά την δυνατότητά τους να γίνουν, να, λειτουργήσουν σε διεθνές περιβάλλον, να ξεφύγουν δηλαδή από το παραδοσιακό εμπορικό τους περιβάλλον. Ε, είδαμε λοιπόν ποιες ε, είναι οι τάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ποιες είναι οι τάσεις αντίστοιχα της διεθνούς αγοράς, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να τις ταυτοποιήσουμε. Μετά το, την εκκίνηση του project αυτού, ε, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κύριο σώμα ενδιαφερομένων Ε, πολλά είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούν να διασταυρωθούν ε, και πολλοί οι φάκελοι οι οποίοι σχετίζονται με το θέμα αυτό. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε δει a few dominate Έχουμε δει, λέω, ότι είναι δυνατόν ε, να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στις εξαγωγικές εταιρείες, ε, οι οποίες ε, βεβαίως εντείνουν τις εξαγωγικές τους δράσεις όταν βρίσκονται σε ένα πιο υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ε, και ε, βεβαίως ε, είδαμε ότι είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να διευρεθούν. Οι δραστηριότητες τους είναι πολλές. Υπάρχει πάντα μια καλή σχέση ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την διεθνή δραστηριοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η σχέση αυτή uh, Η σχέση αυτή ε, ε, ε, είναι πιο έντονη σε μερικές χώρες από ό,τι σε κάποιες άλλες. Αλλά το σημαντικό αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο εδώ είναι το πρώτο στοιχείο. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ε, παραγωγικότητα μπορεί να ε, οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα, θέλουμε να βασιστούμε κυρίως σε αυτό. Uh, uh, Και ε, στα πλαίσια αυτά πρέπει να βασιστούμε στο ανθρώπινο δυναμικό η διεθνής δραστηριοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, βεβαίως είναι ε, βασίζεται σε μια αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων οι οποίες ε, οδηγούνται προς την υψηλή παραγωγικότητα. Υπάρχει διαφοροποίηση και της οικονομικής διάρθρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε την ε, υπόθεση αυτή χρησιμοποιώντας και προηγούμενα στοιχεία και δεδομένα και προσπαθήσαμε να βρούμε ε, την ε, στατιστική σχέση μεταξύ των στοιχείων αυτών τα προηγούμενα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. There are many missing words for key statistics in many countries, so we focus on French small and medium enterprises. Ε, λοιπόν, και στην προκείμενη περίπτωση λοιπόν είδαμε ότι υπάρχει μια τροποποίηση της δομής των επιχειρήσεων ε, κυρίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάνω από 50 ε, ε, εργαζόμενους Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις πρέπει εδώ να ε, συγκριθούν με τις ε, επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στην εσωτερική αγορά και πρέπει να βρεθεί η διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές ε, τις επιχειρήσεις. Πριν σας δώσω τα αποτελέσματα αυτής ε, της ε, έρευνας πρέπει να πω ότι συγκρίναμε τις ημεδαπές, ε, δηλαδή τις εταιρείες οι οποίες έχουν συναλλαγές στην ημεδαπή και αυτές οι οποίες έχουν στην αλλοδαπή και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στον ανθρώπινο δυναμικό και την παραγωγικότητα στις ε, εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ε, δηλαδή βλέποντας ας πούμε το, το ανθρώπινο δυναμικό ε, το, τον, στο, στις διεθνείς επιχειρήσεις έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό ε, ικανοποίησης των εργαζομένων. Και επίσης πρέπει να πω ότι Υπάρχει μεγάλη διάσταση ε, όσον αφορά κυρίως τις υπηρεσίες ανάμεσα στις ε, εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην ΕΜΕΔΑΠΗ και αυτές ε, που λειτουργούν και στην αλλοδαπή. Η διεθνής δραστηριοποίηση τον, ε, ε, ε, έχει σχέση και με το cash flow και με, την, με τους δείκτες, τους οικονομικούς δείκτες οι οποίοι τελικά δείχνουν την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων αυτών. Θα δούμε τώρα κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά δίνοντάς σας τα αποτελέσματα, την έκβαση. κάθε οικονομικός δείκτης δεν είχε σημαντικό ε, συντελεστή ε, σε σχέση με την εσωτερική δραστηριοποίηση. Απ' την άλλη πλευρά, είδαμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια διεθνοποίησης ε, των ε, επιχειρήσεων ε, σε σχέση πάντα με την παραγωγικότητα, με το μέγεθος της εταιρείας και σε σχέση με το αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να έχει στην παρουσία της μικρομεσαίας επιχείρησης η διεθνής της διάσταση. Επίσης, ελέγξαμε την ε, σχέση ανάμεσα την, ανάμεσα στην ε, ε, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και την γενικότερη κατάσταση της αγοράς. Μπορεί να, εκεί βλέπουμε πολλές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Ε, εκεί προκύπτουν διάφορα προβλήματα όσον αφορά ας πούμε τις δασμολογικές επιβαρύνσεις που μπορεί να είναι ψηλότερες ε, σε μια χώρα από ότι σε ε, άλλη χώρα και είναι γεγονός ότι στις χώρες οι οποίες έχουν άρει τις δασμολογικές τους, τα δασμολογικά τους προσκόμματα εκεί είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. πάντως γενικώ δεν βλέπουμε να υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα ε, στα διάφορα στοιχεία αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει εμείς, ε, άμεση επίπτωση της γενικής οικονομικής κατάστασης στη διεθνοποίηση των ε, ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν πιστεύω πάντως ότι τα... Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν παίζουν ρόλο στην διεθνοποίηση ας πούμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επομένως, επιβεβαιώνεται η σχέση ανάμεσα στην Μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ε, παραγωγικότητα και την ε, επενδυτική ένταση αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι ε, ε, παράγοντες που να δυσχεραίνουν τη σχέση αυτή. Η παραγωγικότητα όταν είναι ψηλότερη ε, τότε μπορεί να αυξηθεί και ο εξαγωγικός ρυθμός. Επίσης, γίνεται πιο αποτελεσματική η ε, επίτευξη του στόχου εάν ε, η οικονομική στήριξη είναι στοχευμένη. και η πρόβλεψη των χρηματοπιστωτικών ε, περιορισμών σε συνδυασμό και με την αυξημένη παραγωγικότητα μπορεί να οδηγήσει σε πιο καλά αποτελέσματα. Για εάν θέλουμε να προβλέψουμε καλά το στόχο, θα πρέπει να αναλύσουμε όλα τα στοιχεία. Και ενδεχομένως θα πρέπει να αναθεωρήσει η μικρομεσαία επιχείρηση για κάποιους ε, από τους ενδιάμεσους στόχους της, λαμβάνοντας υπόψη και την γενικότερη κατάσταση του κλάδου. Επίσης να δει κατά πόσον υπάρχουν ειδικές σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κλπ. Πρέπει... Ναι, καταλαβαίνω ότι πρέπει να τελειώσω. Επίσης, η διασφάλιση των πόρων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή με την οποία με ακούσατε. Να είστε καλά. Yeah. Um, σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης βλέποντας τα πράγματα υπάρχουν σαφώς διαφοροποιήσεις για τις ανάγκες και για τη συμμετοχή. Αλλά το ότι ενισχύει την παραγωγικότητα η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι προφανές νομίζω, κάτι το πρόδειλο. Δεύτερο σε πάει Χαίρομαι να καλωσορίσω από την Παγκόσμια Τράπεζα την κυρία Ανδρέα Έγκερ. Χαίρετε. Είναι η εκπρόσωπος της Βρυξέλλες της Παγκόσμιας Τράπεζας και έχει πολύ μεγάλη πείρα στις ε, αναλύσεις ακριβώς ε, αυτών των φαινομένων παγκόσμια. Και θα μας παρουσιάσει τις δικές της απόψεις ε, υπό το δικό της πρίσμα να εξευρεθούν δυνατότητες κεφαλαίων για την παγκοσμιοποίηση προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πνεύμα, στο πρίσμα της παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή για την διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Υπό το πρίσμα μας το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά αυτών που κάνουμε. Και έτσι πάντα παρακολουθούμε με ανησυχία, βλέπουμε με ανησυχία ότι μετά από την κρίση που έπληξε την Ευρώπη βλέπουμε πολλά χρηματοπιστωτικά <clears throat> ιδρύματα να μειώνουν τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα από τα κύρια θέματα είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουν όταν θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε παγκόσμια κλίμακα και χρειάζονται επενδύσεις. Είναι ένα κοινό θέμα για τις ε, ΜΜΕ. Αυτά λοιπόν που θα πω αφορούν τη χρηματοδότηση της επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρωτού πω δύο λόγια ποιοι είμαστε και τι κάνουμε για τις ΜΜΕ, να σας πω από πού προερχόμαστε από τον ιδιωτικό τομέα, από την ε, ακριβώς προοπτική προέλευση της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αγορές. Χρειαζόμαστε, ε, προερχόμαστε από διαφορετική προέλευση από ε, την ε, προοπτική των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων χωρών. Έχουμε μακρά προϊστορία έργου υποστήριξης για μεγάλο όγκο χρηματοδοτήσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 4,5 δίσο όσον αφορά χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Γιατί λοιπόν θα διαρωτάστε να ε, βρισκόμαστε σε μια συζήτηση για την ΕΕ και την χρηματοδότηση των ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε προκλήσεις και κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν είναι τα ίδια είναι κοινά όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες πολύ, μεγάλο μέρος της πείρας μας θα είναι χρήσιμο πιστεύω για αυτή την προσέγγιση. Να σας δώσω με δύο λόγια μια επισκόπηση πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα προσεγγίζοντάς το με τον τρόπο που εργαζόμαστε και αυτή η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιείται και από αυτήν για την πρόσβαση ως ένα από τα στοιχεία κλειδιά να δίνεται άμεση εμπορική χρηματοδότηση, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση συνεργαζόμενη με τις διάφορες τράπεζες και σε επίπεδο συνέργειας και επίσης ε, για τη δημιουργία, την οικοδόμηση χρηματοοικονομικών θεσμικών οργάνων. Θα επανέλθω σε αυτό. Μία από τις κύριε προκλήσεις είναι να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να δανείζουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερη κλίμακα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο και για τις αναδυόμενες αγορές. Αυτό θα το γνωρίζετε και από τη δουλειά μας ε, για τις επενδύσεις ε, υπέρ του ε, κλίματος, θετικού κλίματος επενδύσεων και συμπεριλαμβάνονται τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλο εύρος λοιπόν για να βελτιωθούν τα πράγματα στη δραστηριοποίησή μας αυτή και αυτός είναι ο λόγος ε, για τον οποίο με αυτό το πνεύμα προσεγγίζουμε τα θέματα των ΜΜΕ πράγματα τα οποία κάνουμε εμείς αλλά και που η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνη προσεγγίζει με το ίδιο πνεύμα. Βοηθούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας για τις παγκοσμιοποιημένες αγορές να συνδεθούν με μεγαλύτερες εταιρείες, να μπορούν να εξάγουν και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η ανοικοδόμηση, η δημιουργία δυναμικού. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάρτιση όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, δεξιότητε που πρέπει να αποκτηθούν και ικανότητε για τα στελέχη το τι μπορεί να γίνει τώρα για την συμπερίληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρηματοοικονομικά από τη λέσχη των 20, πώς μπορούν ε, οι παγκόσμιοι διαμορφωτές των οικονομικών πολιτικών να δράσουν. Αυτό είναι κάτι που παντού εξετάζεται γιατί όλοι συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τι μπορεί να γίνει. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, ε, μπορώ να δώσω πολλές πληροφορίες. Θα ήθελα να πω ότι επειδή έχουμε σε βάθος έρευνα που γίνεται εξετάζοντας 164 διαφορετικά πρότυπα χρηματοδότησης ΜΜΕ όσον αφορά τις υπηρεσίες που διαθέτουμε, αυτά τα οποία σας λέω από τη δική μας δουλειά και από την έρευνα όσον αφορά την ε, λέσχη των 20, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η ΜΜΕ και στις ε, αναδυόμενες αγορές και στις ανεπτυγμένες αγορές με, τον, με αυτή την προσέγγιση πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στις περισσότερες χώρες αντι, εκπροσωπούν το, μεγαλύτερο ε, ε, ανθρώπινο δυναμικό σε αριθμούς. Είναι λοιπόν η ραχοκοκαλιά, έχουν το, ε, το κλειδί στα χέρια τους για την ανάπτυξη καινοτομία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης. Η εκμετάλλευση αυτού του δυναμικού θα ήταν κάτι το επωφελές για όλους. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω είναι ότι πέρα από το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν σε όλες τις οικονομίες στη λέσχη των 20 G20, 6% προσελκύουν των επενδύσεων συνολικά και μία από τις προκλήσεις λοιπόν βλέπουμε που διαμορφώνεται σε σχέση με όλα αυτά είναι ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συντριπτική τους πλειοψηφία εξαρτάται από χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τράπεζες για τη χρηματοδότησή τους. Μία από τις ε, μεθόδους που αντιμετωπίζουμε εμείς αυτά τα θέματα και ξέρω ότι υπάρχουν και πολλοί που εμπλέκονται και το αντιμετωπίζουν με παρόμοιο τρόπο τι μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ρόλος των χρηματοοικονομικών ε, ιδρυμάτων τραπεζών για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ. Κάναμε έρευνα βλέποντα τι μπορεί να γίνει, τι γίνεται με τι τράπεζε για να εξυπηρετηθούν, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Και πάλι αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και σε πολλέ ευρωπαϊκέ τράπεζε ω αρχέ. Τράπεζε με τι οποίε συνεργαζόμαστε και εμεί. Ένα από τα θέματα είναι ότι η χαμηλή γνώση, μικρή γνώση που υπάρχει, η ε, έλλειψη ε, πραγματογνωμοσύνης, ε, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το να διαχειριστούν ένα δάνειο προς, σε σχέση με μια μικρομεσαία επιχειρήση, επιχείρηση συνεπάγεται κάποια γραφειοκρατική δαπάνη, κάποια έξοδα, η επιβάρυνση, μέσα στο έργο της Λέσχης των 20 για τις προς, κατα, τους προσανατολισμούς που πρέπει να ακολουθηθούν ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις ε, συγκεκριμένες αρχές που αφορούν και την, τα θέματα αγορών, ιδιαίτερα την ενίσχυση των δυνατοτήτων δυναμικού για τις αγορές, κάτι που μπορεί να υποφελήσει τις ΜΜΕ, αποτελεσματική αρρωγή σε σχέση με τις τράπεζες, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο σε περίοδους κρίσης η δυνατότητα δανειοδότησης και η εμπλοκή και του, ε, ε της σωστής αντιμετώπισης ε, των ΜΜΕ δημιουργώντας ε, δυναμικό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο η πρόσβαση σε κεφάλαια, είναι πολλά περισσότερα συμβουλές και υποστήριξη συνοδευτικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν αποδίονται στο έργο ε, διεθνούς ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές. Και επιπλέον να δούμε αδρές, σε αδρές γραμμές κάποιες γενικότερες ε, ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτών των θεμάτων στη συζήτηση. Το κυριότερο θέμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι είναι διαφορετικέ μεταξύ του οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Διαφοροποιούνται μεταξύ του. δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα και πρέπει να ληφθούν αυτέ οι διαφορέ υπόψη και οι ανάγκε του, έστω και σε αυτό το κλίμα, το, τη, τη μικρή κλίμακα είναι διαφορετικέ πολλέ φορέ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη για ποια μικρομεσαία επιχείρηση μιλάμε. Υπάρχουν μικρέ επιχειρήσει που είναι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορεί να χρειάζονται πολύ στοχοθετικά εξειδικευμένη υποστήριξη από πλευρά τη δράση μα. Δεν θα βοηθήσει μία συνταγή όλες τι επιχειρήσει ε, χωρίς να ληφθούν και άλλα μέτρα πέρα από την χρηματοδότηση. Συμβουλευτική ε, συνδρομή, υποστήριξη, συνοδευτική παρακολούθηση, ε, διευκόλυνση των επαφών τους με τράπεζες κτλ. Δεύτερο στοιχείο, χρηματοπιστωτικά θεσμικά όργανα. Όπως ανέφερα παρακολουθούμε το πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με τράπεζες που δεν παρέχουν δάνεια και πιστώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν οξυνθεί οι όροι του παιχνιδιού και η κρίση. Το πώς μπορούν λοιπόν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα με κοινέ δράσεις, με δημιουργία θεσμών, είναι κάτι που μπορεί να είναι ωφέλιμο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το εξετάζει αυτό. Πρέπει να γίνουν περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήδη θα μπορούσε να διαδραματίσει ε, ε, σπουδαίο ρόλο για να ε, βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Όπως διαφέρουν μεταξύ τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολύ μικρές τέτοιες επιχειρήσεις, υπάρχουν start-ups, επιχειρήσεις που ξεκινούν και δραστηριοποιούνται τώρα εκ του μηδενός και διαφορετική υποστήριξη χρειάζεται ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες, χρηματοοικονομικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για τις διαφορετικές αυτές επιχειρήσεις στην ε, τροχιά τους, στη δράση τους. Ένα άλλο σημείο, ενθάρρυνση της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Είδα, πολλοί πελάτες μας έχουν αυτή την κλίμακα και έχουμε, πρέπει να ενθαρρύνουμε εντός εισαγωγικών μεγάλες επιχειρήσεις να διεθνοποιηθούν και να παγκοσμιοποιηθούν το κάνουμε αυτό σε σχέση με τον τομέα αυτόν στην παγκοσμιοποίηση, βοηθώντας μια εταιρεία να αναπτυχθεί όταν έχουμε μια τέτοια επιχείρηση με πολύ μεγάλη υποστήριξη πίσω τη, μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Α το δούμε αυτό τώρα υπό το πρίσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πόσο πολύ πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για αυτέ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα, να δώσουμε μια χείρα βοηθεία είναι πολύ σημαντικό. Και τέλο θέλω να αναφέρω δύο λόγια για την ε, χρηματοοικονομική κάλυψη ε, των αναγκών από πλευρά του εμπορίου βλέπουμε μεγάλος όγκος κεφαλαίων επενδύεται και χρησιμοποιείται για την χρηματοπιστωτική υποστήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων. Μεγάλο μέρος αυτής της αγοράς καλύπτεται και έχει πριτανεύοντα ρόλο εκεί ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το εμπόριο. Ό,τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε, προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο κενό που πρέπει να καλυφθεί Πρέπει λοιπόν και αυτή είναι η τελευταία μας παράκληση, το τελευταίο μας αίτημα να εξεταστεί, να εξετάσετε την δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης των εμπορικών δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε θερμά. Οι προκλήσεις αυτές πρέπει έτσι να αντιμετωπιστούν. Όχι μόνο σε σχέση με την χρηματοδότηση, αλλά και σε σχέση και με τις συνθήκες πλαισίου που εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον κατάλογο προτεραιοτήτων ώστε συνολικά να έχουμε θετικά αποτελέσματα στο τέλος ως ε, τελευταία έκβαση ως αποτέλεσμα. Χαίρομαι που τώρα μπορώ να ε, καλωσορίσω τον κύριο Έριχ Χουίμερτ που είναι για το Eurocommerce εκπρόσωπος και παρίσταται. Όμως ιδιαίτερα φυσικά και λόγω της πείρας του από το εμπορικό επιμελητήριο Αυστρίας. Το οικονομικό εμπορικό επιμελητήριο σίγουρα και στα άλλα κράτη μπορεί να υφίσταται, αλλά για την Αυστρία υπό το πρίσμα το δικό σας μπορείτε να μας αναφέρετε εσείς το τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε για την πρόκληση για το πλαίσιο αυτό του ε, εμπορικού επιμελητηρίου ε, σε σχέση με την Αυστρία 99% των μελών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, οικονομική και κοινωνική εταίροι στην Αυστρία στον τομέα της χρηματοδότησης προσφέρουμε κυρίως συμβουλευτικές, συμβουλευτική υποστήριξη για τις επιχειρήσεις και για τη δραστηριοποίησή τους στις εξαγωγές αλλά έχουμε και συμβουλευτικό ρόλο και για τις επενδύσεις έχουμε σε 170 χώρες γραφεία εκπροσώπησης και έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις συνολικά που διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στις εξαγωγικές δραστηριότητες στις εξωτερικές αγορές. Οι ε, εμπορικοί ακόλουθοι, όπως τους αποκαλούμε, είναι απεσταλμένοι, είναι εντεταγμένοι σε πρεσβείες της Αυστρίας. Εκεί έχουν θέση και έδρα στην εκάστοτε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντική σημαντικοί πυλώνες και στηρίγματα, υποστήριξη για την οικονομική δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων να προσεγγίσουν και να έχουν πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα όπως προαναφέρθηκε να δραστηριοποιηθούμε όχι μόνο για το θέμα της χρηματοδότησης στην παγκοσμιοποίηση γιατί πρέπει να σκεφτούμε και το πρώτο βήμα. Τι θέλω να κάνω, τι θέλω να εξαγάγω, πού και θέλουμε να προσφέρουμε υποστήριξη ώστε να υποστηρίξουμε συμβουλευτικά τις εξαγωγές. Έχουμε coaches, συμβούλους για τις εξαγωγές στις επιχειρήσεις που διαθέτουν συμβουλευτικά την πείρα τους και οικονομικά μπορούν να συνδράμουν τις επιχειρήσεις αυτές. Και υπάρχει και επιδότηση, κάλυψη του κόστους και των δαπανών, μια de υποστήριξη, μια ελάχιστη σε ελάχιστο επίπεδο υποστήριξη που διασφαλίζεται από πλευράς ε, δικής μας. Τώρα, Αναφέρθηκε ήδη πιο πριν, η κατάσταση για τις επιχειρήσεις δεν είναι καθόλου απλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει επιφύλαξη όταν αντιμετωπίζονται οι ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων επειδή η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση λόγω της ε, κρίσης, πιστοτικής κρίσης και κρίσης χρέους είναι πολύ οξυμένη. Από την άλλη πλευρά είναι πολύ επιφυλακτικές οι τράπεζες. Δεν δίνουν εύκολα δάνεια και πιστώσεις ε, για πολλούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει απαιτούν και εγγυήσεις, όλο και περισσότερες εγγυήσεις οι τράπεζες για να δώσουν δάνεια ή πιστώσεις. Σύντομα λοιπόν, με δύο λόγια, θα είναι η πιο σύντομη παρουσίαση των προτάσεών μας. Προτάσεων που εμείς ασκώντας αυτή τη δραστηριότητα lobbying στο πλαίσιο της Βασιλείας 3, συμφωνιών Βασιλείας 3, χαίρομαι που εσείς ως αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε επιληφθεί αυτού του θέματος και παρακολουθείτε αυτές τις ε, υποθέσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων κεφαλαιακής κάλυψης, κάλυψης με κεφάλαια των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει αυτό να αποτελέσει μια δυνατότητα να δράσουμε για να καλυφθούν οι ανάγκες τους, να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους και να αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τις εμπορικές δραστηριότητες και εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Να αποφύγουμε πλήγματα εις βάρος αυτών των επιχειρήσεων. Και σημαντικό είναι και να δούμε και τις δομές και διαφρόσει των τραπεζών στην Ευρώπη έχουμε πολύ διαφορετικές δομές στο τραπεζικό τομέα. Με μικρές τράπεζες, μεσαίες τράπεζες, μεγαλύτερες τράπεζες ή μεγάλες τράπεζες και όλα αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να βρουν στο λιανικό εμπόριο, για παράδειγμα, εταίρους όπως είναι μικρές ή μεσαίες τράπεζες και τέτοιου είδους σύμπραξη να εξετάσουμε. Τώρα και η ιδέα η διεθνοποίηση να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, να την εκμεταλλευτούμε για να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο εγγυήσεων, ένα ταμείο εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επόμενη χρηματοοικονομική περίοδο προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει. Τα μέσα αυτά, τα χρηματοοικονομικά μέσα να τα ενισχύσει, να υπάρξει η κάλυψη των εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους όσον αφορά τα επιτόκια για τη χορήγηση δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορέσουμε να προαγάγουμε και το ανθρώπινο δυναμικό και υπάρχει και πρόταση για το European Venture Capital από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θα βρίσκεται υποσυζήτηση επίσης και η δυνατότητα χρηματοδότησης από ε, τις ε, ευρωπαϊκές ε, δραστηριότητες, επενδύσεις από, τις δραστηριότητες, από πλευράς της Ευρώπης και ένα εξειδικευμένο θέμα βραχυπρόθεσμη διασφάλιση, εξασφάλιση πιστώσεων για τις εξαγωγές. Και εδώ υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια επιδότηση, ενίσχυση που θα μπορεί να διατίθεται όσον αφορά την διάθεση προϊόντων στις διεθνείς αγορές, στις εξαγωγές δηλαδή από κάποιες επιχειρήσεις. Προβλέπεται Βέβαια η απαγόρευση δημόσιας επιδότησης και υποστήριξης όμως πρέπει να δούμε ποια δυνατότητα θα μπορέσει να δοθεί να υποστηρίξουμε την δραστηριοποίηση στον τομέα των εξαγωγών χωρίς επιδοτήσεις να υπάρξει μια διασφάλιση των πιστώσεων για τις εξαγωγές ή να υπάρχει μια ασφάλεια που θα συνάπτεται για την κάλυψη των εξαγωγικών κινδύνων. Δεν είναι απλά θέματα αυτά. Αυτά εισαγωγικά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ganz herzlichen Dank. Πρόεδρο, Σα ευχαριστούμε θερμά. Είσαστε πολύ εξειδικευμένο όσον αφορά τι ανάγκε για αυτόν τον τομέα, για τι απαιτήσει όσον αφορά το οικονομικό επιμελητήριο, όσον αφορά την ενίσχυση των κεφαλαίων, τη κεφαλαιακής ε, ε, υποστήριξη για τη διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ πάλι είναι σαφής όχι μόνο η άμεση ανάγκη διασφάλισης ε, κονδυλίων, αλλά η διασφάλιση των όρων και των συνθήκων πλαισίου που μπορούν να βοηθήσουν στη διεθνή δράση αυτών των επιχειρήσεων. Τελευταίο τώρα, χαίρομαι που τον Λουκ Χέντριξ, μπορώ να τον καλωσορίσω, τον κύριο Λουκ Χέντριξ ανάμεσά μας, προέρχεται από τον Σύλλογο, την Ένωση για την οποία κάνουμε λόγο την Ένωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τον Σύλλογο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Του δίνω τον λόγο για να μας παρουσιάσει τις απόψεις του για τη διαμόρφωση αυτών των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με προσκάλεσε απόψε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση μαζί σας θέλω να υιοθετήσω μια τελείως άλλη διαφορετική πρόπτικη από εκείνη που υιοθέτησαν οι προλαλήσαντες ε, επαΐοντες. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Στον τίτλο λέγεται «Πρόσβαση σε κεφάλαια για τη διεθνοποίηση». <clears throat> Προσπελασιμότητα, πρόσβαση σε κεφάλαια έχει εγγραφεί στο θεματολόγιο, στην ατζέντα των οργανώσεών μας εδώ και πολλά χρόνια και στα άλλα θεσμικά όργανα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα τα προβλήματα, τα επίκαιρα, επίκαιρα και σημερινά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικά. Και δεν νομίζω ότι εδώ και σήμερα θα βρεθεί η λύση σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Επικεντρωνόμενοι στην παγκοσμιοποίηση και την πρόσβαση στα κεφάλαια, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω και εγώ ότι και εμείς βλέπουμε την παγκοσμιοποίηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και αυτό είναι αυτό που θα έπρεπε διεθνώς να γίνεται. Η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι παραπάνω από τις εξαγωγές. Είναι ένας άλλος τρόπος, ας το πω έτσι, η διεθνοποίηση δεν είναι μόνο οι εισαγωγές αλλά και οι εισαγωγές. Ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων όπως το λιανικό εμπόριο που προσπαθούν όλο και περισσότερο να εισάγουν από τρίτες χώρες για να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η διεθνοποίηση για μας είναι και οι εξαγωγές αλλά και οι εισαγωγές. Και τούτου λεχθέντος αμέσως μπορώ να αναφερθώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο, ρόλ, ο λόγος, ο, ο όρος ΜΜΕ πολλές φορές αποτελεί αντικείμενο κατάχρησης ρώτησε η προλαλή σα, δεν χρειάζεται να υπησέλθουμε σε λεπτομέρειες, 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη, 99 και παραπάνω της 100 είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάμπολες από αυτές είναι επιχειρήσεις ενός ατόμου του ιδίου του επιχειρηματία και συνεισφέρουν για, σε τεράστιο βαθμό για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε μια περίοδο κρίσης είναι οι μόνες οι οποίες συνεχίζουν να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι κανείς σε αυτή την αίθουσα μπορεί να έχει ή έχει αμφιβολίες για τη σπουδαιότητα των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Επανερχόμενος και πάλι στο σημερινό θέμα που μας απασχολεί, ποιες είναι οι δυσκολίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την παγκοσμιοποίηση, οι ενδυνάμει δυσκολίες. Ξέρω ότι όλο και περισσότερο το Ευρωκοινοβούλιο θέλει όλο και περισσότερο βάσεις δεδομένων, που θα βασι... Ε, επιχειρήματα που θα βασίζονται εξειδικευμένα σε βάσεις δεδομένων. Έχουμε και μία μελέτη από τις ε, γαλλικές οργανώσεις για τις ενδυνάμει δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν, πρώτο σημείο και αυτό φυσικά δεν είναι τίποτα το περίεργο και παράξενο, είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας που εξορισμού είναι υπεύθυνο ε, για τις εξαγωγές σε μια τέτοια μικρή επιχείρηση. Ιδιαίτερα η δημιουργία επιπλέον απασχόλησης αποτελεί επιβάρυνση ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που έχουν μέχρι και έξι απασχολούμενους. Δεύτερο πρόβλημα, να εξεύρουν καλά καταρτισμένο προσωπικό να έχουν προσωπικό που να έχει τις αναγκαίες δεξιότητες για τα εμπορικά θέματα. Μπορεί να έχουν στο εθνικό επίπεδο τους αρμόδιους και καλά καταρτισμένους υπαλλήλους, αλλά όχι υποχρεωτικά και για το εξωτερικό εμπόριο και για τις εξαγωγές στο, στην παγκόσμια κλίμακα. Πρέπει λοιπόν να εξευρεθούν αυτοί οι καταρτισμένοι για τα θέματα του διεθνούς εμπορίου. Και μετά η διασφάλιση των κεφαλαίων, της πρόσβασης στα κεφάλαια, η αντιμετώπιση επιπλέον της καθυστέρησης εξοφλήσεων και πληρωμών και η αντιμετώπιση των προϊόντων μαϊμούδων, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά και νομικά μέσα για να προστατευτούν από προϊόντα απομίμησης. Και πάλι λοιπόν η έλλειψη νομικών και οικονομικών μέσων αποτελεί πρόβλημα για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για να υπάρχει μια σε ιδανικό πλαίσιο πολιτική για τις εξαγωγές και και παγκοσμιοποίηση. Όλα αυτά ευθυγραμμίζονται με αυτά που είπε και η κυρία Έγκελ. Οι προσωπικές συμβουλές και οι συνδρομή σχετικά είναι κύρια ανάγκη. Μία θηρίδα που πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη να ενημερώνει και να πληροφορεί. Ένα από τα προβλήματα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν είναι επίσης η έλλειψη γνώσεων, έλλειψη πληροφοριών, στοιχείων και γνώσης που αφορά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εξαγωγές αλλά και όρους και για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού με τις οργανώσεις και ενώσει ε, επιχειρηματιών. Επίση, θέλω να αναφερθώ στην πρόσφατη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά τα θέματα παγκοσμιοποίηση τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εξαιρετική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινά με τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων μέτρων σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο των μέτρων και ρυθμίσεων για τις εξαγωγές. Υπάρχει και υπήρχε τεράστια ανάγκη να γίνει αυτό και έχει ήδη ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το έργο και από κοινού εκπροσώπους των ενώσεων και συλλόγων ε, επιχειρηματιών και επιχειρήσεων. Σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων, όταν έρχεται η στιγμή μια μικρομεσαία επιχείρηση να αποδηθεί στις αγορές, αμέσως αντιμετωπίζουν άμεσα χρηματοοικονομικά προβλήματα ή περιορισμούς, περιορισμούς ε, δυναμικού, προσκόμματα, εμπόδια, ακόμα και γλωσσικά εμπόδια. Διότι ακόμα προτού ξεκινήσουν και όλα τη διεθνή δραστηριοποίησή τους, αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους, το μάρκετινγκ, τις εσωτερικές διεργασίες, ε, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλες αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν χρηματοδότηση και κονδύλια και είναι αρκετά δαπανηρές. Σήμερα, ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει αίτημα για ένα δάνειο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύ συχνά, για να μην πω όλα πάντα, θεωρούνται ως ε, πελάτες υψηλού κινδύνου όταν έχουμε εξαγωγικές δραστηριότητες λοιπόν βλέπουμε ότι σε σχέση με προορισμού σε τρίτες χώρες αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διασφαλίζουν πιστώσεις και δάνεια. Ήδη το ανέφερε η συνάδελφός μου που μίλησε πριν. Το μεγάλο πρόβλημα τούτη τη στιγμή είναι ε, βεβαίως η εφαρμογή των συμφωνιών. Έχουμε και κάποια, κάποιο ε, χαρτί προσανατολισμού όσον αφορά το θέμα αυτό και έχουμε και μια έκθεση η οποία ε, ε, σε σχέση με τη Βασιλεία 3 ε, και έχουμε βεβαίως και κάποιο προβληματισμό όσον αφορά την υλοποίηση της Βασιλείας 3 κυρίως όσον αφορά την χρηματοδότηση ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. In European ε, επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να λαμβάνονται κάποια μέτρα. Πρόσφατα, ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, έδωσε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι κανείς δεν ξέρει εάν τα χρήματα αυτά τελικά φτάνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν όντως τα καρπώνονται τα χρήματα αυτά. Επομένως και εκεί χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ακόμα έτσι ώστε να υλοποιηθεί πραγματικά το, το έργο. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η παγκοσμιοποίηση χρειάζεται, δηλαδή το να γίνει κανείς να, παίξει σε διεθνέ επίπεδο, χρειάζεται, ε, επενδύσεις αλλά στην επένδυση η απόσβεση, η επιστροφή των χρημάτων έρχεται αργότερα ε, και επομένως θα πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί το μέλλον της, ε, της ε, επιχείρησης. Εδώ λοιπόν παρεμβαίνει η δημόσια στήριξη η οποία δεν θα αφορά μονάχα τα οικονομικά χρηματοδοτικά αλλά στήριξη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές καθεαυτές ε, και βεβαίως ε, θα πρέπει η στήριξη να είναι ε, πραγματικά ορισμένη, συγκεκριμένη για ε, τους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεσαίες με από 50-100 υπαλλήλους, κάτω από 50 υπαλλήλους, αλλά επίσης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, συγκεκριμένη δηλαδή ε, ε, στήριξη κυρίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτές που χρειάζονται περισσότερο την βοήθεια. Αλλά βεβαίω μπορούν να δημιουργηθούν και ευρύτερα στοιχεία στήριξη ή προγράμματα στήριξη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Α πούμε, ε, κάτι που σχετίζεται με την οικονομική τους κατάσταση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη, τεράστια ανάγκη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ε, λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο να έχουν καλή πληροφόρηση και επίσης σχετικά με τον τρόπο έγκαιρης και ορθής πληρωμής στις διάφορες χώρες. Ε, η καθυστερημένη πληρωμή είναι τεράστιο πρόβλημα για πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται σε χώρες εκτός της δικής τους, ε, αυτό είναι ένα πολύ ε, οξύ πρόβλημα και εδώ θα περιμέναμε κάποια στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να διευκολυνθούν οι πληρωμές των ε, ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να βρουν τις απαραίτητες κόχες της αγοράς. Δηλαδή, σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και οικονομικά απαγορευτικό για πολλές μικρές επιχειρήσεις ε, να ε, συμμετάσχουν ας πούμε σε κάποια έκθεση, ε, να βρουν πού θα μείνουν, πώς θα... Και ξέρετε τα έξοδα ε, για την συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση είναι ίδια για τη μικρή και τη μεγάλη επιχείρηση. Επίσης το κόσμο είναι βεβαίως ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο στον κανονισμό κόσμο Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ένας τομέας που θα πρέπει να διευρυνθεί περισσότερο. Τελευταίο σημείο, κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε και θα θέλαμε εδώ να αναφερθούμε και στην έκθεση ε, της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής και Κοινωνικής ε, Επιτροπής, ε, μια πρόσφατη έκθεση της ΕΟΚΕ, η οποία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει νέα ε, υποστηρικτικά ε, εργαλεία, ας πούμε ε, εγγυήσεις, διευκόλυνση σε παροχή εγγυητικών επιστολών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ολοκληρώνοντας... Ε, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πάρει κανεί ε, δάνεια. Η τραπεζική πίστη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ε, και βεβαίω η εξωτερική εξέβρεση, μάλλον η εξέβρεση εξωτερική σηματοδότηση είναι τεράστιο πρόβλημα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όσον αφορά τι εκκινήσει, τα startups των επιχειρήσεων, εκεί είναι σχεδόν αδύνατο να πάρει κανεί δάνειο. Από τη στιγμή ε, που οι τράπεζες βλέπουν ε, μία χρονιά ε, που είναι λίγο χειρότερη, τότε κλείνουν τις πρόφυγες του δανεισμού. Είχαμε πολύ κακά παραδείγματα, πολύ ενδεικτικά παραδείγματα μικρών και πολύ μικρών ε, ε, επιχειρήσεων ε, που θέλουν να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά σχήματα. Όλα είναι καλά και στο τέλος βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα προκύπτει στην τράπεζα η οποία αρνείται οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι λοιπόν η πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Οι τράπεζε έχουν κλείσει απολύτω τι τρόφιγγε, δεν δίνουν καθόλου χρήματα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ για το τι κάνουν οι τράπεζες. Ε, θα έχουμε και ακρόση και θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Και εγώ το βλέπω ότι γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ πιστώσεων για καινοτομία ή προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη πλευρά για πιστώσεις που έχουν κάποια σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να προδικάσω τι θα πούν οι ομιλητές. Λέω να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να τοποθετηθεί πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά εσείς αγαπητοί συνάδελφοι θα έχετε σειρά να παρέμβετε. Από την Επιτροπή έχω τη χαρά τον Head of Unit από την Γενική Διεύθυνση Enterprise Επιχειρηματικότητας Επιχειρήσεων ο κύριος Έγκερχαρτ, ο που είναι ε, επί μεγάλο χρονικό διάστημα γνωστός μας για τις δραστηριότητες και τις επαφές που έχουμε μαζί του. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Θα ήθελα απλά να επικεντρωθώ σε δύο σημεία και θέλω να ξεκινήσω με αυτά που είπε ο κύριος Σέντριξ πιο πριν όσον αφορά τα θέματα της ε, ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση διότι είναι σημαντικό πιστεύω ότι ακόμα και το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης είναι η χρηματοοικονομική κάλυψη με κεφάλαια αυτών των αναγκών, πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα που απαιτεί και άλλα μέτρα συμβουλές, υποστήριξη και πληροφορίες και ενημέρωση όσον αφορά τις αγορές τρίτων χωρών για αυτές τις επιχειρήσεις που πρέπει αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στις ΜΜΕ αλλά φυσικά και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα και τα λοιπά για συγκεκριμένα προϊόντα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο στόχος μας είναι απόλυτα σαφής. Λέμε ότι σήμερα 25% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διασυνοριακά δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, διαμεθοριακά, αλλά ακόμα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο 13% ξεπερνούν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολούνται με το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε αυτό το 13% αυτών των ΜΜΕ να μπορέσει να εξομοιωθεί με το υπόλοιπο μέσο όρο. Όμως η προοπτική είναι ανάγκη να το δούμε. Χρειάζεται ως προοπτική να καλύψουμε επιπρόσθετα μέσα μέτρα και δράσεις ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο συσχετίζεται με τις παρατηρήσεις, εισαγωγικές παρατηρήσεις της κυρίας Έγκερ. Είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα, σε αυτή την προοπτική που εμείς υιοθετούμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικά, να δούμε την παγκοσμιοποίηση ως ένα φυσικό μέρος και τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου σφαιρικά. Αυτό τι σημαίνει, ότι πολλά από τα θέματα τα οποία συσχετίζονται με την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών <clears throat> είναι φυσικά και τα μακροπρόθεσμα θέματα. Έχουμε και τα βραχυπρόθεσμα βέβαια, αλλά σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο, σε ένα μακροπρόθεσμο ε, χρονορίζοντα, πρέπει να δούμε αυτή την ανάγκη και όπως είπαν πολλοί ομιλητές, ξέρουμε ότι έχουμε κρίση αυτή τη στιγμή, μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε και οι υπηρεσίες που εμείς ε, είμαστε υπεύθυνοι για το έργο αυτό δεν μας δίνουν κάποια ένδειξη ότι θα υπάρξει κάποια βελτίωση. Η κατάσταση είναι λοιπόν δυσχερής, δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να το δούμε σε ένα πλαίσιο γενικότερο και σφαιρικό. Να δούμε τα μέσα και εργαλεία που χρειάζονται και που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δοθεί υποστήριξη και να χρηματοδοτηθούν οι ΜΜΕ. Και έχουμε και το πρόγραμμα για την ε, Competitiveness and Innovation Program, CIP, SIP, πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούμε, αλλά κατά το τέλος του προγράμματος θα έχουμε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις που θα καλύπτουμε. Και μεγάλο ποσοστό από αυτές τις επιχειρήσεις είναι μικροεπιχειρήσεις. Οι μικροεπιχειρήσεις είναι ξεχωριστές σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο, αλλά και στις μελέτες που έχουν συνταχθεί και αναφέρθηκαν και εδώ και άλλες μελέτες έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά λοιπόν, χαρακτηριστικά και ανάγκες όσον αφορά την χρηματοδότησή τους και την παγκοσμιοποιημένη τους δραστηριοποίηση. Επιπρόσθετα πέρα από το σύστημα εγγυήσεων πιστώσεων έχουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ε, δάνεια και πιστώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την διασφάλιση κινδύνων στις αγορές, ε, κεφαλαιακές αγορές ε, χορήγησης κεφαλαίων κινδύνου, ε, και πρέπει να δούμε σε σχέση με αυτή την περίοδο οικοδομώντας, ε, δημιουργώντας πάνω στην πύρα που έχουμε συλλέξει σε αυτή τη χρονική φάση εργαζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα νέο πρόγραμμα για την επόμενη περίοδο, το πρόγραμμα COSME, το οποίο ακολουθεί άρρηκτα και δίνει συνέχεια στις προηγούμενες δράσεις. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα που αφορά το πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 για την χρηματοδότηση των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάνοντας λόγο για την έρευνα και ανάπτυξη σχετικά είναι σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό ότι υπάρχει σαφής ένδειξη και αναφορά ότι καινοτόμες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται έννοια κλίμακα επειδή ασχολούνται με ένα τέτοιο τομέα και προϊόν που ε, μπορούν ας το πω σε, σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο να το διαθέσουν Τούτων λεχθέντων πρόεδρε, πιστεύω ότι όλοι μας θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε και να κάνουμε χρήση των προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και συζητούμε. Να τα δούμε ως ένα στοιχείο, ως ένα σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και δραστηριοποίησης παγκόσμια αυτών των επιχειρήσεων. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ θερμά και δίνω τώρα τον λόγο στους συναδέλφους. <clears throat> Εσείς έχετε πρώτος τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. πάρα πολύ σύντομο. Πρώτα απ' όλα να σας πω ποιο είμαι. Πολύ σύντομα. Τζον. Από το πιο μικρό νησί του Μεσογείου, της Μεσογείου που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι από τη Μάλτα δηλαδή. Και ε, παραπάνω από το 1 πέμπτο του προϋπολογισμού, μα του ΑΕΠ μας, συγγνώμη, προέρχεται από την βιομηχανία και όχι από, την, τον τουρισμό, όπως νομίζει κανείς. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, εμείς δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε εσωτερική αγορά. Το περισσότερο μέρος της βιομηχανίας καλύπτεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, εγώ ήμουν υπουργός... Ε, βιομηχανίας και είδα το πρόβλημα ανάποδα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ότι έπρεπε να δω ε, τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ας πούμε, ε, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε για μικρομεσές, για μη μία ε. Το πρόβλημα είναι ε, το, το πρόβλημα των startups, των ε, ε, επιχειρήσεων που ξεκινούν. Ε, απ' την άλλη πλευρά έχουν τα προβλήματα των επιχειρήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Επομένως μπορεί να βρούμε ας πούμε κάποια κοινά στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά έχουν και πολλές ιδιαιτερότητες. Επίσης δεν είναι το ίδιο πράγμα να ψάχνει για χρηματοδότηση μια εταιρεία, μια επιχείρηση η οποία έχει 149 εργαζόμενους και άλλο μια που έχει έναν ή κανέναν ή μόνο τον ιδιοκτήτη. Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα ε, υπάρχει όσον αφορά με τις τράπεζες, αλλά είναι ε, παρεμπίπτον. Μάλλον τα, τα, τα παρεμπίπτοντα δηλαδή δεν μπορούν να, να παρασχεθούν από τις τράπεζες, μεταξύ άλλων η ασφάλεια, οι εγγυήσει. That usually industrial estates are Επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες μας έχουν ε, ε, οικοδομηθεί σε κρατική γη, σε δημόσια γη. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες, αλλά εμείς ε, φτάσαμε σε διαφωνίες όσον αφορά το τι εννοεί ο καθένας λέγοντας long lease agreement, συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης. Ε, ε, και αυτό είναι ας πούμε ένα παρεμπίπτον ε, μεγάλο ζήτημα, δηλαδή η χρήση της γης, ποια, ποια είναι η γη και μην ξεχνούμε ότι η γη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εγγυητικό στοιχείο για την παροχή δανείων. Η τράπεζα δεν πρέπει να δανείσει αν δεν έχει δύο ασφαλίσεις. Άρα ξαναερχόμαστε στην αρχή του κύκλου ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ε, η τράπεζα αλλά τα παρεμπίπτοντα που δίνει η τραπεζική ε, πίστη. Πρέπει να δούμε τα περισσότερο τις τρομερές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, οι, οι κινήσεις επιχειρήσεων στα startups ε, και επίσης ε, την δυσκολία που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την καινοτομία, ας πούμε, τη χρήση της καινοτομίας, τη χρήση της δημιουργίας. Βάζουμε όλα, όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές τις εταιρείε σε αυτό το καζάνι ε, το, στο οποίο βάζουμε προμετωπίδα μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ η κάθε μία από αυτές έχουν διαφορετικά προβλήματα, έχει διαφορετικά προβλήματα. Πρέπει να δούμε το κάθε ένα είδος με άλλο μάτι, από άλλη οπτική γωνία. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι το ίδιο να έχεις δύο εργαζόμενους και 102. Δεν είναι το ίδιο 15 εργαζόμενοι με 150 ή 250. Ε, γι' αυτό λοιπόν εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν ο, βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να τις δούμε ξεχωριστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού ο εισηγητή λάβει αμέσω τον λόγο, εγώ ίδιο έχω εγγραφεί στον κατάλογο αγορητών. Ενέγραψα τον εαυτό μου. Και θα ήθελα του πραγματογνώμενου επαείοντε να του ρωτήσω κάτι. Αφενό, ποιο είναι ο ρόλο ουσιαστικά των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών θεσμικών οργάνων. Ακούστηκε κάπω ότι η Ευρωπαϊκή λέει, Τράπεζα Επενδύσεων έχει κάποιο ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα 37 εκατομμύρια όμως δεν είναι σαφές αν φτάνουν σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως αποδέκτες. Πόσο υψηλός θα έπρεπε να είναι ο όγκος αυτός χρηματοοικονομικά για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, μια και με αυτή την κρίση θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τι πρέπει να γίνει ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά να μπορούν να κάνουν χρήση να απολάβουν αυτών των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ιδιαίτερα όσο αφορά τις προτάσεις υπέρ αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, τι γίνεται ουσιαστικά με τα διαθροτικά ταμεία. Συζητάμε για 370 δισεκατομμύρια ευρώ των διαθροτικών ταμείων ως κονδύλια. Και πρόκειται για κέντρο βάρους, με την ε, καινοτομία ως κέντρο βάρους δεν μπορούν τα διαθωτικά αυτά κονδύλια να χρησιμοποιηθούν περισσότερο για την διάθεση κονδυλίων για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης, να επισκέπτονται κάποιες εκθέσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να διευκολύνονται οι όροι και οι συνθήκες πλαίσιο που έχουν, πλαισίου που έχουν για τη δραστηριοποίησή τους. Και τρίτον, σε σχέση με τις τράπεζες αναφέρθηκε ότι υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με Συμφωνία Βασιλείας 3, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας υπάρχει διαφορετική αντίληψη όσον αφορά τις πιστώσεις που θα μπορούσαν να, να εγκρίνονται. Η δική μου πείρα είναι ότι πιστώσεις για μέτρα φιλοπεριβαλλοντικά στη Γερμανία για παράδειγμα εγκρίνονται και διατίθενται. Εντάξει, πιστώσεις και κονδύλια για την ε, παγκοσμιοποίηση όμως λιγότερο, σε μικρότερο πλαίσιο. Τρεις ερωτήσεις προς τους επαΐοντες. Και τώρα θα δώσω τον λόγο λοιπόν στον εισηγητή. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρία λόγια να πω. Έχουμε λοιπόν την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας την οποία ε, για την οποία είμαι υπεύθυνο όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να δράσουν σε διεθνές περιβάλλον. Ακούσαμε πολλά πράγματα σήμερα. Ακούσαμε επίσης εμπειρογνώμονες με διαφορετικό βαθμό ή θέση τεχνογνωσίας. Είχαμε δύο εκπροσώπους από δύο πολύ ισχυρούς ε, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς. European level and another organized και έχουμε ε, και άλλες ε, ακούσαμε και εθνικές ας πούμε απόψεις από το αυστριακό επιμελητήριο π.χ. Ε, νομίζω ότι περισσότερα από αυτά τα οποία είπαν συμπλήρωναν το ένα το άλλο και νομίζω ότι μπορούμε να απομονώσουμε τρεις περιοχές προβλημάτων ε, και στη δομημένη μας συζήτηση θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτές τις τρεις ενότητες προβλημάτων, τα clusters των προβλημάτων. Κατά την άποψή μου, η πρώτη δέσμη προβλημάτων, η πρώτη ομάδα προβλημάτων εγγύεται στο θεσμικό πλαίσιο Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε το κλίμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δούμε ας πούμε το κατά πόσον θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει κάποιο νέο εργαλείο όσον αφορά το δανεισμό, όσον αφορά ε, τις εξαγωγικές διαδικασίες κτλ. Επίσης, όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά τα λειτουργικά του ε, έξοδα κτλ. Δεύτερη ομάδα προβλημάτων, ε, τα κανονιστικά και νομικά βήματα τα οποία πρέπει να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας πούμε, τι είδους ε, τέτοια βήματα ε, μπορούμε να τους ε, συστήσουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως, δηλαδή στα παρεμπίπτοντα, στην πίστη, την τραπεζική. Σωστά είπε ο συνάδελφος μπροστά όλα αυτά που είπε γιατί αν θέλουμε βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξουν άλλα κίνητρα, άλλα ε, ε, μέτρα ε, υποστήριξης έτσι ώστε ας πούμε να μειωθεί το, το, το πρόβλημα, το χάσμα του δανεισμού, κυρίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι τρεις κύριες ομάδες προβλημάτων που απομόνωσα εγώ. Με ικανοποίηση πρέπει να πω ότι βλέπω ότι έστω και σε αυτήν την πολύ ε, ε, πρώτη έτσι, φάση συγγραφής ε, της έκθεσής μου είχα την στήριξη μέσω των ιδεών που μας παρήχαν οι καλεσμένοι μας εμπειρογνώμονες. Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι γεγονός ότι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι ίδιες όμως, για να διευκολυνθούν τα πράγματα, εγώ θα, θα επιλέξω μάλλον να μην εντείνω ακόμα περισσότερο αυτήν την ε, ασάφεια των ορισμών Ξέρουμε νομίζω όλοι όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τι ε, εννοούμε. Ξέρουμε τι είναι μικρομεσαία και τι δεν είναι ακριβώς μικρομεσαία επιχείρηση. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τον τεχνικό ορισμό για χάρη ευκολίας γιατί θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα και δεν το θέλουμε αυτό. Αυτά. Και εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ ενθαρρυντικά και πολύ ανανεωτικά τα όσα ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω τον λόγο πάλι στους τέσσερις επαΐοντες. Ακούσατε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούσατε και κάποιες ερωτήσεις από ευρωβουλευτές. Σας καλώ τώρα να τοποθετηθείτε και να απαντήσετε. Ο κύριος Γιούτο, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά, δεν έχω κάποια καλή δεδομένη άποψη για το καλύτερο τον καλύτερο τρόπο επίλυσης των χρηματοοικονομικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε σχέση και με το workshop finance εξετάζοντας τις ανάγκες, τα αποτελέσματα από αυτή την πλευρά η χρηματοοικονομική δομή, η δομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Και όπως είπε και ο κύριος Χέντριξ, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν συλλογικά με τον ίδιο τρόπο, συλλήβδιν. Πρέπει οι ανάγκες τους να λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά και ειδικά εξειδικευμένα. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη χρονική στιγμή να γίνεται αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Έγκελ. Um, um, ευχαριστώ για τον ρόλο των IFIs ε, που μπορούν να έχουν ε, οι μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα δεδομένης της κρίσης και η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε κεφάλαια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύει τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι έτοιμη και μπορεί να συμμετάσχει. Οι δυνατότητες και τα μέσα που έχει με εγγυήσει μέσω των τραπεζών, τη δραστηριοποίηση κεφαλαίων κινδύνου, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ήδη. Επίσης, δεν είμαι σίγουρη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά ό,τι μπορεί να γίνει σε σχέση με συμβουλές και συνδρομή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με τράπεζες είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και η αύξηση του κεφαλαίου για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση ως πρόταση. Πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν αν γινόταν αυτό, αν αυξανόταν το κεφάλαιο και σε προηγούμενη φάση διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των αναγκών των επιχειρήσεων και για τις τράπεζες και τα δάνεια για την ε, παγκοσμιοποίηση θα ήθελα να αναφέρω ότι για τράπεζες που δανείζουν κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πελάτες υψηλού κινδύνου αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Οτιδήποτε θα μπορούσε λοιπόν να γίνει για την είσοδο στις διεθνείς αγορές αυτών των επιχειρήσεων, αυτό τον κίνδυνο θα τον κάνει όπως τον θεωρούν οι τράπεζες ακόμα μεγαλύτερο για τις τράπεζες. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέσο διευκόλυνσης εισαγωγών-εξαγωγών. Δεν έχω κάποιες έτοιμες απόψεις κομμένες και ραμμένες για, την, για ένα τέτοιο μέσο. Έχει αναφερθεί όμως Πιστεύω ότι υπάρχουν θεσμοί και δυνατότητες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εγχείρημα η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χαρτογραφήσει το τοπίο και μετά να καλυφθεί με κάποια πρόταση το, εκείνο που απουσιάζει, εκείνο που χρειάζεται και πρέπει να καλυφθεί ως ανάγκη είναι μια δεδομένη δυνατότητα. Θα μπορούσε να ενδυναμώσει το μπορούν να γνωρίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι κάποιο τέτοιο μέσο υπάρχει. Επίσης, ε, συντάσσονται και εκθέσεις ε, για επιχειρήσεις και καταδεικνύεται ότι ετήσια θα μπορούσαν πολλά περισσότερα να γίνονται για να βελτιωθεί το γενικότερο περιβάλλον, η ατμόσφαιρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην, στην Ευρώπη. Παρατηρήσεις και σχόλια από δική μας πλευράς που θα μπορούσαν έτσι να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Ο επόμενος αγορητής ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στην ίδια την Αυστρία μάλλον περιορισμένη εμβέλειας η σημασίας διότι υπάρχει ε, επαρκές εύρος μέτρων και δυνατοτήτων στην Αυστρία και σε σχέση με την Ευρωζώνη. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι οι ασφάλειες, εχέγγυα, εγγυήσεις χωρίσεις δανείων και πιστώσεων. Υπάρχουν αρκετά τέτοια μέσα. Κάλυψη αυτών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι πολύ μεγάλη δυνατότητα και από εθνικούς θεσμούς ε, με την αντασφάλιση για παράδειγμα που παρέχεται όσον αφορά επενδυτικά ταμεία. Είναι ένα καλό μέσο αυτό που μπορεί να επεκταθεί ακόμα περισσότερο η χρήση του. Η ιδέα ότι θα μπορεί να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό ταμείο εγγύσεων είναι θετική. Υπάρχουν πολλά μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ωστόσο και σε σχέση με το ΣΥΠ στον ορίζοντα 2020 με τα μέτρα που έχουμε και τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει τα χρηματοοικονομικά αυτά μέσα ως θεσμούς να τα ενισχύσει περισσότερο ώστε να υπάρχει πιο ενεργός ρόλος ε, και να δούμε πώς μπορούν αυτά να δράσουν για πιστώσεις και δάνεια που θα μπορούν να διευκολύνονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ε, δυνατότητα, δηλαδή κάλυψη κινδύνου όχι μόνο άμεσα σε σχέση με το δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και ανακυκλούμενη. Αυτό είναι το προτέρημα έναντι των επιδοτήσεων ή ενισχύσεων. Για τα διαθροτικά ταμεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 11 προτεραιότητες. Η μία είναι η καινοτομία, η άλλη είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το κέντρο βάρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μία προτεραιότητα επενδυτική προβλέπεται για νέα πρότυπα επιχειρήσεων για τη διεθνοποίηση. Αυτό έχει εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το θέμα των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια, ε, ποιες πιστώσεις ε, θα πρέπει να μπορούν να εξεταστούν θα πρέπει να δούμε λιγότερο το για πιο χρονικό διάστημα, αλλά και το θέμα του rating, η φερεγγιότητα όσον αφορά τη ρευστότητα, διαδραματίζει και αυτή ένα ρόλο. Και το θέμα της δυνατότητας μέσω αυτής της φερεγγιότητας να καταλήξει κανείς σε κάποια πίστοση. Υπάρχουν και εθνικά μέσα που πρέπει να εξεταστεί αν επαρκούν για αυτές τις ανάγκες. Δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά ε, να θέτει ένα αίτημα στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο μια επιχείρηση. Πρέπει πρώτα να στρέφει στρέφεται στις εθνικές δομές και στους εθνικούς θεσμούς, παρότι αποτελεί άλλο θέμα τώρα το θέμα της αντασφάλισης. Να σκεφτεί κανείς ε, για παράδειγμα την εθνική ε, εγγύηση για τέτοιες ε, εξαγωγικές δραστηριότητες, αν καλύπτει τους κινδύνους και τις ανάγκες ή χρειάζεται ένα άλλο πρότυπο. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ. Πέτρος, ευχαριστώ. Και τελευταίος, ο κύριος Χέντριξ θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως να απαντήσουμε πρώτα στη δικιά σας ερώτηση. Μήπως θα μπορούσε ο μιλητής να βάλει λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά του. Δεν ακούμε καλά. Ε, είναι πολύ μακριά. Ευχαριστούμε. Ε, σχετικά με την ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ναι, είναι γεγονό ότι εγώ αναφέρθηκα στα 30 εκατομμύρια, τα οποία δεν ξέρουμε ε, πώ θα δοθούν, πού θα δοθούν, με ποιο τρόπο. Ε, και δεν ξέρουμε πού θα πάνε τα περισσότερα χρήματα και πού τα λιγόμενα. Επίσης ε, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτησή σας ακριβώς. Εσείς είπατε ότι θα πρέπει τα χρήματα να φτάσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχετε κάποια πρόταση Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τεχνοκράτης, λέει ο κύριος Χέντριξ, δεν έχω ε, την ε, απάντηση, δεν, δεν ε, είμαι εμπειρογνώμονας τεχνοκράτης σχετικά με το θέμα αυτό. ξέρω ότι... Πρέπει κάτι να γίνει για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση. Όσον αφορά τα διαφορετικά ταμεία τώρα, ξέρω ότι ε, θα πρέπει να γίνει ε, μια προσπάθεια έτσι ώστε τα, στα, τα διευθυντικά ταμεία να μην γίνουν μια κολυμβήθρα όπου θα μπαίνουν όλα τα προγράμματα και οποιοδήποτε προβληματικός ε, τομέας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τα διορθωτικά ταμεία να χρησιμοποιηθούν για το λόγο για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί ε, και βεβαίως είναι πολλές ε, οι ανάγκες μικρών επιχειρήσεων που δεν ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα. Όσον αφορά τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολλή συζήτηση έγινε. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε ο ε, βουλευτής ε, από τη Μάλτα. Είναι γεγονός ότι ο καθένας έχει άλλες ανάγκες. Δεν μπορεί κανείς ε, να συγκρίνει μία πολύ μικρή επιχείρηση με ένα-δύο εργαζόμενους και μία άλλη που θεωρείται πάλι μικρομεσαία αλλά έχει 249 εργαζόμενους. Θέλει άλλη τεχνογνωσία, άλλη αντιμετώπιση κτλ. ο παρόν ορισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει, είναι ελληματικός, έχει υποστεί πολύ, πολλές επικρίσεις. Είναι σαφές πάντως ότι θα πρέπει, ακόμα και όταν μιλάμε για μη μη ε, να διαφοροποιούμε τις μικρές και τις μεγαλύτερες μεταξύ αυτών η κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, micro enterprises, ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, διότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης <coughs> όσον ε, αφορά αυτές τις micro enterprises. Τέλος, πιστεύουμε ότι η χρηματική στήριξη ή οποιαδήποτε άλλη στήριξη θα πρέπει να αφορά α, τις επιχειρήσεις οι οποίες περισσότερο χρειάζονται τη στήριξη αυτή και αναφέραμε πάντα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά μπορώ να επαναλάβω το ίδιο. Το πρόσφατο ανακοινοθέν το οποίο αφορά τις ε, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, θέλουν να μεγαλώσουν είναι πάρα πολύ ε, θετική ανακοίνωση και νομίζω ότι εδώ η Κομισιόν έλεβε υπόψη της στα σχόλια των εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε και με την Ένωση των Επιχειρήσεων Business Organization αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό Ευχαριστούμε πολύ κυρία Έγκερ. Θέλετε να λάβετε τον λόγο και πάλι παρακαλώ. Uh, σύντομα, Πρόεδρε, ναι, ευχαριστώ. Απλά και μόνο ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το οποίο αναφέρθηκε όταν γίνεται λόγος για νέα θεσμικά όργανα όσον αφορά τη χρηματοοικονομική υποστήριξη εξαγωγών. Πιστεύω ότι ως προτέρημα το βλέπουμε ότι ουσιαστικά σε όλα τα κράτη-μέλη έχουμε θεσμικά όργανα σε σχέση με αυτή τη δραστηριοποίηση θα έλεγα ας χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας προτού δημιουργήσουμε νέα. Φυσικά το θέμα της κρατικής ενίσχυσης ή ε, επιχορήγησης είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη αν θα χρειαστεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές ή όχι. Αλλά είναι ένα εξειδικευμένο θέμα και όχι ένα θέμα δημιουργίας ξεχωριστού θεσμού. Δεύτερο, όταν έχουμε το θέμα, όταν γίνεται συζήτηση όπως την ερώτησή σας για πιστώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων όπως το βλέπουμε έχει καλό έλεγχο της χρήσης γιατί υπάρχει και κίνητρο που έχει ενταχθεί στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των επιμέρους τραπεζών. Αλλά φυσικά μπορούν τα πράγματα να ίσως και να βελτιωθούν περαιτέρω και με μεγάλο ενδιαφέρον θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή τη δυνατότητα να υπάρχει μια καλύτερη ε, ε, ε, διευρυμένη δυνατότητα οι τράπεζες έτσι να συμμετάσχουν και θα ήθελα να σχολιάσω και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή έχουμε εξωτερικούς επαΐοντες που ασχολούνται με αυτό. Συμφωνούμε με τους επαΐοντες που ανέφεραν ότι δίνει ένα ολόκληρο φάσμα, ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων όταν έχουμε το σχεδιασμό, θέμα σχεδιασμού ε, ειδικών μέσων για ειδικέ κατηγορίε, πρέπει έτσι να το δούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, εσεί θέλετε να πείτε δύο λόγια. Πάρα πολύ σύντομα ε, να ευχαριστήσω τους ε, εμπειρογνώμονε και βεβαίω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Ε, ήταν ανανεωτικές οι ιδέες που άκουσα, ε, ήταν, θα αποτελέσουν και πηγή έμπνευσης για την ε, έκθεσή μου και βεβαίως μου δίνουν και κάποια καλά επιχειρήματα και κάποια στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσω στην έκθεσή μου. Να ευχαριστήσω φυσικά και την γραμματεία για μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια της ημέρας σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητά. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πραγματογνώμονες για άλλη μια φορά, να τους ευχαριστήσω θερμά. Κάνατε τον κόπο να έρθετε εδώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να συζητήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Ευχαριστούμε και τη Γραμματεία για τη διοργάνωση αυτή τη ακρόαση. Και πάλι προ του επαΐοντες θα ήθελα να πω ότι πάντα τίνουμε δίκο ους ευήκο αότα στα όσα έχετε να μας πείτε και ο εισηγητής και οι άλλοι ευρωβουλευτές. Αν έχετε κάποιες ιδέες ή απόψεις πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε κεφάλαια για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στείλτε μας την, την ιδέα σας ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Διακόπτουμε τώρα τη συνεδρίαση μέχρι τις 6, 18.00. Μετά ο Επίτροπος Ντεχούχτε θα κάνει μια τοποθέτηση από πλευράς του. Ευχαριστώ. σε beta Good, liebe Kolleginnen und Πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, χαιρετίζω όλους σας και πάλι για άλλη μια φορά για το τελευταίο αυτό τμήμα της συνεδρίασής μας, συνεδρίασής μας απόψε, όπως είχαμε συμφωνήσει. Και τώρα έχουμε ευκαιρία να έχουμε μια δήλωση από τον Επίτροπό μας, κύριο Ντεχούχτ, για την ΑΚΤΑ. Και θα έχουμε μετά και όπως έχει συμφωνηθεί από τις πολιτικές ομάδες, μία τοποθέτηση από εκπρόσωπο ευρωβουλευτή να ή ευρωβουλευτή από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, κύριε Επίτροπε, εσείς πρώτος, παρακαλώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ, σε αυτή τη ε, στιγμή των κρίσιμων αποφάσεων. Αύριο πρέπει να ε, ληφθεί μια απόφαση η οποία αφενός αφορά τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες και ε, κατά το άλλο της τμήμα αφορά την ίδια την ουσία του πράγματος. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ε, γνωμοδότηση από την ε, ε, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να δει εάν οι κανονισμοί σχετικά με την παραχάραξη και την απομίμηση συμμορφούνται προς και συνδυάζονται με την Χάρτα Θεμελιωδών Ελευθεριών. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος όσον αφορά το θέμα αυτό. Η άκτα, όπως είπα και προηγουμένως, θέλει να προστατέψει τους ανθρώπους και όχι να αποτελέσει πρόβλημα για οποιοδήποτε, ε, με οποιοδήποτε τρόπο. Υπάρχει επίσης και η εσωτερική μας νομοθεσία, η λεγόμενη κοινωνικό και, κοινοτικό και ακή κομινοτέρα ε, και θα διευρυνθεί το κεκτημένο αυτό αύριο. Αλλά οτιδήποτε είναι σήμερα παράνομο θα ε, εξακολουθήσει να γίνει και αύριο παράνομο και μετά την κύρωση της ε, άκτα. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες ε, ε, πρέπει σωστά να ερμηνευθούν. Γι' αυτό ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αύριο ένα μέρος της αυριανής απόφασης θα αφορά το κατά πόσον η συμπερίληψη της άκτα στην διακυβερνητική συμφωνία ήταν σωστή. Επίσης θα πρέπει να συμφωνηθεί το τι θα γίνει μετά από την ε, συνεκτίμηση όλων των δεδομένων από το Συμβούλιο και μετά τη γνωμοδότηση ε, του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εμείς δεν θέλουμε gouvernement de juge, όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστή ερμηνεία των θεμελιωδών ελευθεριών, ερμηνεία την οποία μονάχα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να κάνει. Ήδη ε, πέρσι είχε ζητηθεί πάλι μέσω προδικαστικού ερωτήματος ε, ε, μια παρόμοια γνωμοδότηση για την άκτα. Τα ζητήματα όμως εξακολουθούν να παραμένουν. Το άλλο τμήμα της επιλογής σας αφορά την ίδια την συμφωνία και το περιεχόμενό της. Η ενδυνάμωση λοιπόν των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ε, δικαιοσύνης και ιδιοκτησία, συγγνώμη. Ε, αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση και επομένως στα πλαίσια αυτά της κρίσης, αυτής της κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε εταιρείε οι οποίες προσπαθούν να προχωρήσουν βάσει των πνευματικών δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεκτιμήσετε και το σημάδι, το μήνυμα που θα στείλουμε στον υπόλοιπο κόσμο μέσω της αυριανής ψηφοφορίας. Αξιότιμα μέλη, Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία από πλευρά σας, ε, εγώ βρίσκομαι εδώ για να σας ε, ε, σταθώ. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε, παρόλα αυτά θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την παρούσα διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου γιατί έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει. Μία αρνητική ψηφοφορία δεν θα σταματήσει τις διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εάν συμμορφούνται οι αποφάσεις, ε, τότε θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όμως, περιμένω ότι ε, το δικαστήριο θα θεωρήσει την άκτα ε, πλήρως συμμορφούμενη προς τις συνθήκες. Επομένως, μπορούν να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, θα μπορούσα να προτείνω κάποιες αποσαφηνήσεις επί της άκτα. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ενδυνάμωση του ψηφιακού περιβάλλοντος. Θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα αυτό υπό το φως των νομοθετικών προτάσεων που έχει αποφασίσει να προβάλλει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν το Συμβούλιο ή μπορεί να αποσαφινιστεί περαιτέρω η μπορει να αποσαφενιστει περαιτερω η εννοια του commercial scale. Επίσης, είμαι ανοιχτό σε συζήτηση για το ε, τι σημαίνει μοίρασμα πληροφοριών ε, στα πλαίσια της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει λοιπόν μια νέα πρόκληση όσον αφορά την κλασική προσέγγιση των δικαιωμάτων πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Όμως δεν έχει συζητηθεί το θέμα βάσει του βασικού δικαίου αυτοί είναι πολύ σημαντικοί λόγοι ε, που μας οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω σκέψης ε, και αποσαφήνισης όσον αφορά το μέλλον του, συστήματος, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης, όταν θα έχουμε ταυτοποιήσει και συζητήσει τις ε, ε οποιασδήποτε δυνατές αποσαφηνίσεις, τότε θα ζητήσω ξανά την γνώμη του Κοινοβουλίου. Ε, εσείς θα αποφασίσετε λοιπόν τελικά πώς θέλετε να κινηθείτε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι όλοι σεβόμαστε την ατομική ελευθερία. Όμως πιστεύουμε ότι η ελευθερία χρειάζεται πλαίσιο και σε μια ε, διαφοροποιημένη κοινωνία δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η ε, απόλυτη ε, ελευθερία. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ελπίζω ότι όλα αυτά θα τα έχετε κατά νου την ώρα της ε, ψηφοφορίας σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε σας θερμά κύριε Πίτροπε για, αυτή, για αυτό το σαφές μήνυμα που μας δώσατε. Όπως συμφωνήσαμε τώρα οι κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου θα έχουν δυνατότητα να τοποθετηθούν, να αντιδράσουν από πλευρά τους. Έχουμε μέχρι τις 6,5 χρόνο μην εξαντλήσετε στο και στο χρόνο παρέμβασή σας για να έχουν όλοι δυνατότητα να παρέμβουν λοιπόν. Από το ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Έχει πρώτη τον λόγο. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Υπάρχουν ανησυχίες ε, και μελήματα σχετικά. Όλοι έχουν αντιληφθεί αυτό το θέμα μέχρι σήμερα, σίγουρα. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπραξε αρκετά ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς αυτές οι ανησυχίες. Σας άκουσα προσεκτικά και με ικανοποιεί ότι είσαστε πρόθυμος, πρόθυμοι να εξετάσετε αυτά τα προβλήματα. Έλπιζα όμως και ευελπιστούσα ότι θα είχαν γίνει όλα αυτά νωρίτερα και θα είχαν συζητηθεί και αποσαφινιστεί. Εδώ βρισκόμαστε όμως σήμερα. Αύριο θα ψηφίσουμε το θέμα της άκτα προς έγκριση και τίθεται το θέμα να το απορρίξουμε κάθετα ή να υπάρξει χρόνος που θα δοθεί. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο στην παρατήρησή σας υπό το πρίσμα ότι θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή τη χρονική στιγμή να πούμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συνενέσουμε ενώ εκρεμεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, η δική μου τροπολογία που κατέθεσα θα την αποσύρω. Δεν μπορώ να την υπερψηφίσω, διότι με την αποσαφήνιση που είπατε εσείς, που ε, δεν έχει ακόμα διασφαλιστεί. Όμως αυτό σημαίνει ότι η λογική απάντηση ήταν να απορρίψουμε την άκτα. Διότι απορρίπτοντα την άκτα, εντάξει, ωραία, θα έδινε κάποια ανακούφιση σε πολλά μέλη διότι για ανησυχίε για τα συνεπαγόμενα. Όμω πιστεύω ότι όλοι μα είμαστε αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών μα, με μία κύρια ευθύνη εδώ. Και αυτό είναι να εκπροσωπούμε του πολίτε μα και τα συμφέροντά του και να αντιμετωπίζουμε τα συνεπαγόμενα προβλήματα των προϊόντων, απομίμηση. Έτσι δεν είναι. Για όλου αυτού τους λόγους λοιπόν πιστεύω ότι η καλύτερη λύση θα ήταν το να ψηφίσουμε υπέρ της αναβολής, να αναβληθεί η ψηφοφορία, να αναμείνουμε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να ακούσουμε τι θα πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το χρόνο που θα υπάρξει ώστε να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών και ημών των εκπροσώπων των πολιτών. Αυτό θα ήταν η καλύτερη δυνατότητα, να μην σκοτώσουμε, δολοφονήσουμε τον ασθενή προσπαθώντας να τον θεραπεύσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το σαφές μήνυμα της σαφή σας τοποθέτηση και ευχαριστώ για το ότι είσαστε και σύντομο στη χρήση του χρόνου. Οι σοσιαλδημοκράτες στη συνέχεια εκπροσωπούνται από τον David Μάρτιν. Παρακαλώ. Yes, in the name of... Μάλιστα, εξ ονόματος της σοσιαλιστικής ομάδας και όχι τόσο συζήτης. Πρώτα απ' όλα να αποσαφινιστεί ότι η ομάδα ως ομάδα, οι σοσιαλιστές δεν ασκούν επικρίσεις στους στόχους της άκτα. Το δεχόμαστε, το ότι έχουμε καθήκον να υπερασπιζόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των Ευρωπαίων δημιουργών και παραγωγών και ότι και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό. Όμως απορρίπτουμε το κείμενο ως πρόταση της άκτα, της συμφωνίας αυτής. Ακούσαμε τα επιχειρήματα και έχουν αναφερθεί πολλές φορές. Θα ήθελα κάποια κύρια ε, στοιχεία να αναφέρω. Πρώτον, πιστεύουμε εμείς ότι η άκτα εσκεμένα ή για άλλους λόγους επιβάλλει μια αστυνομική δύναμη που θα παρεμβαίνει, θα επεμβαίνει στο διαδίκτυο. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Δεύτερον, ανησυχούμε και η Επιτροπή το αναγνωρίζει αυτό ότι ο ορισμός των εμπορικών ζητημάτων και δεξιοτήτων στη συμφωνία αυτή δεν καθορίζεται επαρκώς και γι' αυτό μπορεί αυτό να είναι επικίνδυνο. Και τρίτον, οι κυρώσεις που προβλέπονται ή εξετάζονται από την άκτα για την κατάχρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι αναλογικές κυρώσεις. Γι' αυτό απορρίπτουμε για όλους αυτούς τους λόγους την άκτα. Τίθεται το ερώτημα να καθυστερήσουμε την ψήφιση για να ακούσουμε ποια θα είναι η νομολογία του Ευρωδικαστηρίου πιστεύω ότι αληθεύει α, έχοντας ε, το ΕΛΚ ε, που ε, σε σχέση με την τοποθέτησή του για την άκτα, τι θα έπρεπε να γίνει για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα πολιτικά δικαιώματα, αν είναι κανείς υπέρ. Αν όμως είναι κανείς κατά της άκτα, δεν βλέπω λόγο να αναμείνει κανείς την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μόνο καθυστέρηση θα βλέπαμε στην αναβολή μιας πολιτικής επιλογής και σε σχέση με την πολιτική επιλογή, η πολιτική επιλογή της ομάδας μας είναι να απορρίψει την άκτα και να γίνει γοργά να ακολουθηθούν οι διαδικασίες και να αναλυφθεί πρωτοβουλία για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συμφερόντων της Ευρώπης από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οι φιλελεύθεροι λίγο αργότερα θα παρέμβουν. Οι πράσινοι τώρα θα έχουν τον λόγο. Thank you. Um... Ευχαριστώ πολύ. Αληθεύει ότι η πράτη ζήτησαν απόφαση του ε, δικαστηρίου και ότι οι συζητήσεις είναι ακόμα ε, ανοιχτές. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα στηριχτεί η άποψη της διαιτησίας για το θέμα αυτό. Και βεβαίως το προδικαστικό ερώτημα το οποίο έθεσε η Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικοστήριο είναι γενικόλογο και ασαφές. Ε, και σε γενικές γραμμές ε, πρέπει να πω ότι συμφωνούμε με αυτό που είπε ο κύριος Μάρτιν ε, και βεβαίως είναι εξαιρετικά αγχωτικό το γεγονός ότι μας αφήνει μόνους μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουμε αυτή την τόσο σημαντική απόφαση. Βεβαίως από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι εμείς πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε δικές μας αποφάσεις μέσω δημοκρατικών διαδικασιών. Από την άλλη μεριά θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο Φένγελ και θα πω ότι όντως θα πρέπει να, δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές έχουν τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που είσαστε παρόν σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. <clears throat> Και όλοι λέμε ότι έχουμε επαφές και είχαμε παρεμβάσει από τους ε, πολίτες μας, ε, emails, ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνήματα και τα περισσότερα ήταν από ανθρώπου από την εκλογική μου περιφέρεια, αλλά είχα και ηλεκτρονικά μηνύματα και από άλλε πλευρέ που έλεγαν ότι είναι ζωτική σημασία για την βιομηχανία, την επιχείρησή του, και σε σχέση με όσου ε, συμμετέχουν σε αυτέ τι επιχειρήσει να υπερψηφίσουμε και έχουμε και άλλου που πιστεύουν ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου αν υπερψηφίζαμε τη συμφωνία αυτή υπό αυτού του όρου τη διαβουλεύση πρέπει να βρούμε κάποιο νόημα στη θέση που πρέπει να υιοθετήσουμε. Πολλοί από εμάς ε, είχαμε συζητήσεις ε, και εξετάσει και είχαμε διατυπώσει ερωτήσεις προς την Επιτροπή και εγώ έχω υποβάλει ερωτήσεις κοινέ και ατομικές προς την Επιτροπή. Αντανακλούν όλα αυτά τις ανησυχίες για την εκπροσώπηση των ε, μηνυμάτων των πολιτών μας που μας διαβίβασαν και που είπαν ότι πρέπει αυτά να σας διαβιβάσουμε. Γι' αυτό πήραμε χρόνο λοιπόν, ασχοληθήκαμε με αυτά και κατά κάποιο τρόπο θλίβομαι για το γεγονός ότι θα αποσυρθούν οι τροπολογίες ε, ε, ε, του ΕΛΚ όσον αφορά την υπερψήφιση. Όμως είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε ποια θα είναι η άποψη δεν, το, του δικαστηρίου. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να βιαστούμε να καταποντιστεί αυτή η συμφωνία. Πρέπει να δούμε τα μελήματα και ανησυχίες των μελών αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής όπως είπαν και άλλοι καλύπτονται ή όχι. Είδαμε όλες τις ομάδες που είπαν ότι ήθελαν να, αναφερθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αναμένουμε τώρα. Αναμένουμε την τελική απόφαση, στο τέρμα πριν από το πέναλτι. Και σε σχέση τώρα με την τροπολογία να αναβληθεί η απόφαση μέχρι ότου υπάρξει το, η ανομολογία του Ευρωδικαστηρίου, να είμαι απόλυτα σαφής. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζω επαρκώς ε, αν ε, οι ανησυχίες μου αυτές όσον αφορά τις ε, τα θέματα εμπορικής κλίμακας μπορούν να ικανοποιηθούν. Δεν γνωρίζω τώρα αν αυτό θα μπορεί να γίνει μέσω μιας ομάδας επέμβασης αστυνομικής δύναμης στο διαδίκτυο και να δούμε το πόσο όλα αυτά θα μπορέσουν να ερμηνευθούν και σε σχέση με τις, ε, τα νομοθετικά πλαίσια και τις συνθήκες. Δεν μπορεί να επιβληθεί όμως από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο ή από έναν ε, προσυπογράφοντα στον άλλον. Γι' αυτό για να είμαστε λογικοί θα λέγαμε παρακαλούμε να υπεψηφιστεί η τροπολογία μας, να υπεψηφίσουμε για αναβολή, δεν υπάρχει ε, βιασύνη να ληφθεί κάποια απόφαση και αν υπάρξουν αβεβαιότητε για την ομολογία, εκείνοι που θέλουν να την καταψηφίσουν μπορεί ίσως να ακούσουν κάτι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που μπορεί να βοηθήσει τα επιχειρήματά τους. Ε, και τότε θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε, να δούμε, θα εγκρίνουμε ή όχι, ή θα καταψηφίσουμε ως Κοινοβούλιο αυτή τη συμφωνία. Δεν υπάρχει διασύνη θα έλεγα. Θα ζητούσα από τους μου να καθυστερήσουν τη λήψη απόφαση μέχρι ότου υπάρξει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Να μην βιαστούμε. Σίγουρα ένα από του λόγου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ανέφερε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό το θέμα το παρέπεμψε εκεί ήταν ότι υπήρχαν πολλά αιτήματα από τους ε, ψηφοφόρους μας, από τους πολίτες μας, ε, από τους ε, βουλευτές. Εμείς ασκήσαμε τα δικαιώματα και τις εξουσίες μας και το καταστήσαμε σαφές ότι έπρεπε να παραπευθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να αναμείνουμε την απόφασή του. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Οι φιλελεύθεροι είναι τώρα σε θέση να παρέμβουν. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η ομάδα μου είχε τη θέση το ότι το Κοινοβούλιο με τη σειρά του θα έπρεπε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θέλαμε να το διαρθρώσουμε με πολλές ερωτήσεις, πολύ ευρύτερες από αυτές τις οποίες διατύπωσε η Κομισιόν. Εμείς όμως ψηφίσαμε ως Επιτροπή και χάσαμε έναντι της πρότασής μας. Θεωρώ ότι το να περιμένουμε να ψηφίσουμε την έκθεση Μάρτιν ανάλογα με τις προσδοκίες της κοινή γνώμης έναντι των ατέλειωτων συζητήσεων που είχαμε για το θέμα τόσο σε επιτροπές όσο και σε ολομέλειες. Και αναγνωρίζω στην Επιτροπή ότι συνεργάστηκε, που μας ενημέρωσε και δεν παραπονεθήκαμε ποτέ για έλλειψη διαφάνειας από την Κομισιόν. Μπάση περιπτώσει όμως σήμερα γνωρίζουμε πάρα πολλά στοιχεία. Και Και θεωρώ, αν κρίνουμε και από το επίπεδο ρημότητας πια της συζήτησης, ότι το να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου θα ξεκαθαρίσουμε κάποιες, άλλες, κάποιες παραπάνω πλευρές. Αυτό θα μπορούσε και να ερμηνευτεί ως πράξη αδυναμίας εκ μέρους του Κοινοβουλίου και έλλειψη οράματος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να λύσουμε πια αυτό το πρόβλημα και γνωρίζοντας και τη θέση των σχεδόν εισηγητών της ομάδας μου στις άλλες επιτροπές, η θέση που συζητήσαμε σε διάφορες συνεδριάσεις μέσα στην Άλτε. Ε, έχουμε ορίσει και μια συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Άλτε, εγώ θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη πλέον αύριο να εκφραστούμε υπέρ της, ε, στην, επί της ουσίας της έκθεσης Μάρτιν. Ευχαριστώ. Η Ενωτική Αριστερά θα λάβει τώρα τον λόγο. Η Γκουε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ για να εκφράσετε την άποψή σας. Εάν υπάρχει κάτι θετικό ε, γιατί σχετικά με την άκτα είναι ότι ανακοίνησε έτσι μια μεγάλη συζήτηση, δημόσια συζήτηση. Και τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο υποκίνησε τη μεγάλη δημόσια συζήτηση, απαιτώντα στην ουσία ε, αυτό αυτή τη συζήτηση και ε, ε, κάνοντας θέμα το περιεχόμενο της ε, συμφωνίας αυτής. Τώρα βεβαίως πρέπει να δούμε την ώρα της νίκης των πολλών, των πολυάριθμων εθελοντών που δούλεψαν για την άκτα και που θέλησαν να ξεπεράσουν ένα πρόβλημα που άπτεται της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Στην αυριανή ψηφοφορία τα μέλη του Κοινοβουλίου της ομάδας μου της νοτικής Αριστεράς θα εκφράσουν την πλειοψηφία των ε, πολιτών ε, το περιεχόμενο της άκτα δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ε, την ε, περαιτέρω ανάλυση κάποιων παραγράφων. Είναι ώρα από τεχνοκράτες ή από δικαστές. Είναι ώρα για πολιτικές αποφάσεις και για πολιτικές προσεγγίσεις. Επομένως, κατά της ε, ε, κατά της ε, ε, ρυθμιστικής παρέμβασης που δεν χρειάζεται σε αυτό το επίπεδο. Η ΑΚΤΑ ήταν μια προσπάθεια των λίγων να ασκήσουν πίεση και έλεγχο κατά των πολλών. Είναι καλό πάντως που σας έχουμε εδώ κύριε Επίτροπε και θα ήθελα να ε, και είπατε κι εσείς ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή ε, η αμφιλεγόμενη συζήτηση. Και εγώ το ίδιο λέω, θα πρέπει να κληθούν οι συνάδελφοι αύριο να καταψηφίσουν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις των πολιτικών ομάδων για την δήλωση, την ανακοίνωση του Επιτρόπου που έκανε πιο πριν και σύμφωνα με τα όσα συμφωνήσαμε ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ όλους, όλες και όλους και μπορούν οι συνάδελφοι την εικόνα για το τι θα κάνουν αύριο να αποφασίσουν τα σχετικά και με τις συζητήσεις στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Ελπίζω ότι μπορούμε αύριο να έχουμε μια υπεύθυνη απόφαση που θα μπορέσουμε να λάβουμε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο.